Colleagues, shall we start? Good afternoon. Καλό σας απόγευμα. Να καλωσορίσουμε και τον εισηγητή. It's Lisbon Day. Congratulations. Colleagues, shall we all sit down? Συνάδελφοι, καθίστε δηλαδή να τελειώσετε με τα πηγαδάκια ή να μεταφερθούν έξω τα πηγαδάκια, ό,τι θέλετε. Um, uh, Πριν συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη, θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που συμφωνήσαμε το πρωί. Αν θέλουμε να έχουμε ουσιαστική συζήτηση αύριο το πρωί για την θέση σε ισχύ της ε, συνθήκης της Λισαβόνα, SWIFT και PNR, χρειαζόμαστε ένα μνημόνιο, ένα επόμνημα από την νομική υπηρεσία για την ε, νομική κατάσταση, για το νομικό υπόβαθρο. Το ζητάμε τελευταία στιγμή, αλλά η νομική υπηρεσία γνωρίζει την κατάσταση και θα μας ε, δώσουν ένα υπόμνημα, τουλάχιστον στα αγγλικά, απόψε, για να προετοιμαστούμε για την αυριανή συζήτηση. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει κάποιος από την νομική υπηρεσία εδώ. Νομίζετε ότι μπορείτε να μας δώσετε ένα τέτοιο υπόμνημα. Θα το διαβιβάσω διότι αντικαθιστώ το, το μέλος της νομικής υπηρεσίας, τουλάχιστον να είναι ενημερωμένη. Ωραία, σας ευχαριστούμε. Ας συνεχίσουμε λοιπόν με τα σημεία 6 και 7 της ημερήσιας διάταξης. Όχι λέει, α μάλιστα 6 και 7 διορθώνει η Πρόεδρος για τις θεωρήσεις μακράς διαμονής και καταχωρήσει στο σύστημα πληροφοριών Σέγγεν και κυκλοφορία των προσώπων με θεώρηση μακράς διαμονής. Ο κύριος Κουέλιου θα μας ε, κάνει μία εισήγηση για τις θεωρήσεις ε, μακράς διαμονής. Έγινε μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων στο 15 Οκτωβρίου και από όσο γνωρίζω ο κύριος Κοέλιο συνεργάστηκε με τους Σκιώδης στο μεταξύ. Η θέση σε ισχύ σημαίνει ότι το πακέτο εντάσσεται στη συναπόφαση. Κύριε Κοέλιο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Όπως ε, είπατε, είχαμε μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων, άρα δεν θα ήθελα να επανέλθω σε όσα συζητήθηκαν. Θα ήθελα να υπενθυμίσω τα βασικά σημεία μόνο. Στις 5 Απριλίου του επόμενου έτους θα τεθεί σε εφαρμογή αυτό το σύστημα το οποίο θα ακυρώσει τις θεωρήσεις C και D. Υπάρχουν όμως περιορισμοί για αυτούς που κατέχουν θεωρήσει μακράς διαμονής μέχρι τότε. Όπως ε, είπαμε, τα κράτη-μέλη θα πρέπει ε, τάχιστα να ε, κατανείμουν, να διανύμουν τις ε, άδειες παραμονής, αλλά εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα επί του θέματος. Άρα Αν θέλουμε να επιλύσουμε αυτή τη λίστα πρέπει να βρούμε μία δεύτερη λύση. Γι' αυτό χαιρόμαστε για την υπόδειξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιλύσουμε το θέμα έτσι ώστε οι κάτοχοι των θεωρήσεων μακράς διαμονής, μακράς διαρκείας να έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας στο χώρο Σέγγεν. Στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων ανέφερα την περίπτωση ενός πολίτη ο οποίος σπουδάζει στο Βέλγιο, έχει μία θεώρηση μακράς διαρκείας αλλά δεν έχει δικαίωμα να μεταβεί στην Ολλανδία να επισκεφθεί μία βιβλιοθήκη και να κάνει μία έρευνα για το διδακτορικό του ή δεν μπορεί να φύγει ένα Σαββατοκύριακο στη Βαρκελόνη για αναψυχή καθαρά. Η διαδικασία αυτή λύγει τον επόμενο Απρίλιο. Εν πάση περιπτώσει, στο μεταξύ, ε, αυτό το φυσικό πρόσωπο δεν έχει δυνατότητα μετακίνησης εντός του χώρου Σέγγεν. Η Επιτροπή μας έδωσε ορισμένε εναλλακτικέ και έτσι συνέταξα και την έκθεσή μου. Θα ήθελα να τονίσω το θέμα της ασφάλειας, διότι η ελεύθερη κυκλοφορία στους κατόχους θεωρήσεων ε, δεν σημαίνει ότι δεν, μάλλον, δεν σημαίνει ότι διακυβεύεται η ασφάλεια μέσα στα πλαίσια αυτών των θεωρήσεων. Στο ΣΥΣ, στο σύστημα πληροφοριών Σέγγεν, θα γίνει ένα check-in έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ως προς το καθεστώς ασφάλειας. Δηλαδή, οι κάτοχοι θεωρήσεων από τρίτες χώρες φτάνουν στα σύνορά μας και δεν μπορούν να τα διαβούν εάν δεν έχουμε πληροφορίες από το σύστημα, εσωτερικό σύστημα Σέγγιν, από το ΣΥΣ. Επρόκειτο για κάτι το παράλογο, γιατί με την τροποποίηση που προτείνουμε θέτουμε ένα προγενέστερο κριτήριο για την ε, καταχώρηση αυτή. Όπως υπενθύμησε και η Πρόεδρος, η θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας θα αλλάξει κάπως την κατάσταση. Φαίνεται ότι θα έχουμε συναπόφαση και στους δύο τομείς, διότι στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα το όλο καθεστώς δεν έχει νόημα. Ως προς θεωρήσεις μακράς διαρκείας θα έχουμε δύο διαφορετικές νομικές βάσεις. Γι' αυτό και παρουσίασα δύο εκθέσεις. Δεν ξέρουμε την ανακοίνωση Omnibus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν ξέρουμε τι θα κάνει με αυτές τις πρωτοβουλίες. Θα ήθελα η Επιτροπή να μας παρουσιάσει αυτή την ανακοίνωση Omnibus το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε να ορίσουμε το νέο νομικό πλαίσιο. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να τηρήσουμε την ε, περίοδο των 8 ε, εβδομάδων για την ακρόαση με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Γι' αυτό προτείνω ένα χρονοδιάγραμμα που να τηρεί τις 8 εβδομάδες και προτείνω την ε, υποβολή τροπολογιών 10 μέρες μετά τη λήξη της περίοδου των 8 εβδομάδων. Όπως σας είπα, τον Απρίλιο του 2010 θα τεθεί σε εφαρμογή αυτό το καθεστώς. Διαφορετικά θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους κατόχους θεωρήσεων μακράς διαρκείας ως προς την θεώρηση τύπου δίκεση. Θα ήθελα να πω ότι η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας είναι πολύ καλή και, εν πάση περιπτώσει, ως προς τις τροπολογίες θα ήθελα να ε, προτείνω στην ΛΥΜΠΕ να δεχτεί τις τροπολογίες της νομικής επιτροπής εκτός από την τροπολογία υπαριθμών 1, διότι θέλει να συμπεριλάβει βιομετρικά στοιχεία στις θεωρήσεις μακράς διαρκείας. Εδώ υπάρχουν ε, δύο προβλήματα, ένα τεχνικής υφής και άλλο ένα ουσίας. Οι θεωρήσεις μακράς διαρκείας εισαγάγονται μέσω ενός στίκερ που δεν μπορεί να συμπεριλάβει βιομετρικά στοιχεία, αλλά δεν έχουμε και αρμοδιότητες να αποφασίσουμε για κάτι τέτοιο η ε, έκδοση θεωρήσεων είναι εθνικό θέμα, άρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να ορίσει πώς τα κράτη-μέλη θα προβούν σε αυτή την έκδοση θεωρήσεων. Άρα δεν έχει νόημα να μπούμε σε μία συζήτηση της τροπολογίας 1 της Νομικής Επιτροπής σε σχέση με τα βιομετρικά στοιχεία, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είναι θέμα δικής μας αρμοδιότητας, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε και προτείνω να μην ακολουθήσουμε αυτή τη συμβουλή για τους λόγους που προανέφερα. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε πλέον το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Νομίζω, έτσι το ερμηνεύω εγώ τουλάχιστον, μιλάτε για τις κινήσεις της νομικής υπηρεσίας αλλά δείτε μάλλον την ε, Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Ναι, ναι, ναι, γιατί σε κάποιε φορέ δεν καταλαβαίνόμαστε. Είναι που έχουμε τόσε υπηρεσίες και τόσε επιτροπές, λέει η Πρόεδρος, και μπερδευόμαστε. Να, καλέσω λοιπόν τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει πρώτη. Είτε ο κύριος Ντεκόστερ, είτε η κυρία Ρετανάγκη. Η Προεδρία όπου να είναι καταφτάνει. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή χαίρεται για, τις, ε, για την ε, προαγωγή των εκθέσεων του κυρίου Κοέλιο. Τώρα στα πλαίσια της συναπόφασης θα ενταχθούν και αυτές οι δύο εκθέσεις. Επίσης ε, τόνισε τη σπουδή που θα πρέπει να μας διακατέχει, διότι στα πλαίσια των θεωρήσεων D και C, η διαδικασία αυτή δεν θα ισχύει από τις 5 Απριλίου του 2010, τότε δηλαδή που θα υπάρξει ο κώδικας θεωρήσεων, θα πρέπει λοιπόν να εξεύρουμε μία λύση. Χαιρόμαστε λοιπόν για την έκθεση του, για τις εκθέσεις του, γιατί υπάρχει σύγκληση απόψεων με βάση τις εργασίες μέχρι τούδε εργασία στο Συμβούλιο και νομίζω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι μπορούμε να εξεύρουμε μια συμφωνία μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Η νομική μας υπηρεσία μας είπε ότι οι οκτώ εβδομάδες διαβούλευσης με τα Εθνικά Κοινοβούλια ισχύουν ακόμα και σε περίπτωση προτάσεων που υποβλήθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Υπάρχει μόνο ένα σχέδιο τροποποίησης μάλλον τροπολογίαση πρόκειται για την τέταρτη τροπολογία που αφορά το επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σχέση με τις διαβουλεύσεις στα πλαίσια του στήματος πληροφοριών Σέγγεν. Η βασική μας ιδέα είναι ο κάτοχος της θεώρησης D να έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως ισχύουν στους κατόχους άδεια παραμονής χωρίς να αλλάξουμε την ουσία ε, αυτών των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κατανοώ την ανησυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς την προστασία δεδομένων, αλλά προβλέψαμε μία τροπολογία που ζητά από τα κράτη-μέλη να τηρήσουν τις προδιαγραφές ως προς την προστασία δεδομένων σε σχέση με το ΣΥΣ 1, προδιαγραφές που αποφασίζονται στο μεταξύ για το SES2 αλλά που δεν έχουν τεθεί σε ισχύ. Θα πρέπει λοιπόν από νομικής απόψεως να το κάνουμε αυτό, μπορούμε να το κάνουμε, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και ορισμένες επιφυλάξεις που υπάρχουν επί του θέματος. Ως προς το θέμα των βιομετρικών δεδομένων, όταν είχαμε μία πρώτη συζήτηση επί του θέματος, θεωρήσαμε ως Επιτροπή ότι το θέμα, η ουσία δεν είναι να θέσουμε βιομετρικά στοιχεία στις θεωρήσεις ΔΕΛΤΑ. Είναι ένα θέμα που θα εξετάσουμε και θα δούμε κατά πώς θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν θεωρούμε ότι διακυβεύεται η ασφάλεια εάν δεν εισαγάγουμε βιομετρικά στοιχεία στη θεώρηση ΔΕΛΤΑ. Ο κ. Κουέλιο μίλησε για τα τεχνικά προβλήματα που υφίστανται όταν ε, εισαγάγουμε τσιπάκια στα στίκερς του διαβατηρίου. Πολλές φορές είναι ε, αδύνατον να αναγνωστούν τα διάφορα μικροτσιπάκια και γι' αυτό ε, υπάρχουν προβλήματα, μπορούν να ανακύψουν προβλήματα για τους ταξιδιώτες. Γι' αυτό συμμεριζόμαστε τις επιφυλάξεις που εξέφρασε ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω, έχει καταφτάσει η Προεδρία στο μεταξύ. Κάποιον βλέπω να σηκώνει το χέρι του. Ποιο θα μιλήσει λοιπόν εξ ονόματο τη Προεδρία. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ανεκάρπορα ονομάζομαι και δυστυχώ, ο συνάδελφο που είναι υπεύθυνο για το θέμα αυτό βρίσκεται στη συνεδρίαση στο Συμβούλιο. Δυστυχώ, λοιπόν δεν θα μπορέσω να σα κάνω σχετική παρουσίαση. Θα τη ωστόσο ό,τι μηνύματα έχετε να μου δώσετε και θα σα. Ε, Ευχαριστώ, λέει η Θα ήθελα να κάνω μία πρόταση. Θα μπορούσε η Γραμματεία να φροντίσει τα ερωτήματα που θα ανακύψουν στην δίχως άλλος πολύ ζωντανή συζήτηση που θα ακολουθήσει να μεταφερθούν γραπτά στο συνάδελφό σας και να μας απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα η Προεδρία. Εντάξει. Ωραία. Ποιος θέλει το λόγο, η κυρία Λάτφορντ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλώ εκ μέρους της κυρίας Μπίκστρομ, η οποία δεν μπορεί να είναι εδώ στην αίθουσα σήμερα. Και θα ήθελα λοιπόν τις δικές της απόψεις να αποδώσω. Πρώτο σχόλιο, το οποίο και συμμερίζομαι, είναι ότι συμφωνούμε με τον Κοέλιο, ο οποίος θεωρούμε έκανε εξαιρετική δουλειά για την έκθεση αυτή. Υποστηρίζει επίση η συνάδελφο τι τροπολογίε που υπέβαλε ο κ. Κοέλιο, Συμπεριλαμβανομένη στις τροπολογίε για τα πρότυπα για την προστασία των δεδομένων και θα πρέπει να ισχύει αυτό και να ορίζεται στα σχετικά εργαλεία. Έχω μόνο το σχέδιο της γνωμοδότησης της κυρίας Μπίκστρομ για την Επιτροπή νομικών υποθέσεων. Δεν έχω τις τροπολογίες και εσείς αναφερθήκατε στις τροπολογίες που θα υποβληθούν για τη γνωμοδότηση αυτή σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τα βιομετρικά στοιχεία. Άρα είμαι λίγο σε μειονεκτική θέση. Δεν τα έχω αυτά. Καταλαβαίνω ωστόσο τι εννοείται για τις πρακτικές δυσκολίες που ανακύπτουν σε ό,τι αφορά τα βιομετρικά στοιχεία στις βάσεις δεδομένων. Δεν τα γνωρίζουν πολύ αυτό το θέμα αυτό όπω ο κ. Κοέλιο. Εγώ ξέρω λίγα πράγματα, αλλά όχι πάρα πολλά. Συμφωνώ ιδιαίτερα με την γενικότερη κατεύθυνση του αιτιολογικού σημειώματος της έκθεσης του κυρίου Κοέλιο, με την οποία συμφωνεί και η συνάδελφός μου. Ο κ. Κοέλιο είναι λίγο πιο διπλωματικός από ότι συνάδελφος. Είναι όντως απαράδεκτο οι πίκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι νόμιμα διαμένουν σε μια χώρα και μπορούν να το αποδείξουν, δεν έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας μέσα στην Ένωση, το οποίο θα έπρεπε να έχουν λόγω διοικητικής ανικανότητα σε ό,τι αφορά άδειε παραμονή. 20 χρόνια μετά από τη σύμβαση σε αυτό είναι απαράδεκτο και το όλο σκηνικό σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία πρέπει να πω ότι είναι απαράδεκτο. Η τροπολογία 38 του 2004 για την ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων πολιτών τα κατοχυρώνει αυτά. γιατί οι θεωρήσεις ε, μακράς ε, διαμονής ε, έχουν λιγότερα περιθώρια, λιγότερα δικαιώματα από ότι οι θεωρήσεις ε, σύντομης διάρκειας. Είναι πραγματικά απαράδεκτο αυτό από τα κράτη-μέλη. Η κυρία Βίξτρομ έχει την αίσθηση ότι θα άρμοζε να ξεκινήσει η Επιτροπή κάποιες μεμονωμένες διαδικασίες επί παραβάση. Γιατί στον πυρήνα των υποθέσεων αυτών είναι τελικά η αποτυχία, η ανικανότητα των κρατών μελών να εφαρμόσουν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αν, έπρεπε, αν έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν, δηλαδή να εκδώσουν εντός των υποχρεωτικών χρονικών πλαισίων της άδεια παραμονής, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν η κυρία Βίξτρομ καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις μεμονωμένες ε, καταστάσεις που επικρατούν στα διάφορα κράτη-μέλη και να κοιτάξει πού χρειάζεται να ξεκινήσουν διαδικασίες επί παραβάση. Υπενθυμίζει επίσης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να στριχτεί στην μακρά μεμολογία, σύμφωνα με την οποία ακόμα και ίσονος ε, σημασίας ε, διοικητικές ε, κακές πρακτικές θα πρέπει να τιμωρηθούν στην περίπτωση που είναι επαναλαμβανόμενες και συνεχιζόμενες. Μπορεί δηλαδή κάθε, ε, τέτοια, κάθε τέτοιο παράπτωμα να είναι ασήμαντο, αλλά επειδή υπάρχει αυτή η συνέχεια, παρόλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν μέτρα και επειδή υποτίθεται ότι τα μέτρα έχουν επίσημα εφαρμοστεί από τα κρατημέλια και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν κενά, υπάρχει άγνοια στα στους αξιωματούχους των Υπουργείων, των Εθνικών Αρχών. Πολύ απλά δεν ξέρουν λοιπόν τι πρέπει να κάνουν. Άρα νομίζω ότι αυτό που θέλει να πει η κυρία Βίξτρομ είναι ότι αυτό δεν σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν τη νομική υποχρέωση να εκδώσουν άδειες παραμονής. Γιατί τελικά τα κράτη-μέλη είναι αυτά που δεν κάνουν αυτό που θα έπρεπε να κάνουν. Πρέπει να υπάρχει πολιτική ορθότητα Κατά τα άλλα, υποστηρίζει όλα όσα είπε ο εισηγητής. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Γιώτοβα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια κι εγώ σαν σκιώδης εισηγήτρια. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την δουλειά που έχει κάνει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κόλλιε και ε, μπορούμε να περιμένουμε μια συμφωνία μέσα στα πλαίσια της πρώτης ανάγνωσης διότι ούτως ή άλλως θα τεθεί σε ισχύ και ο, κωδικό, και ο κώδικας για την, για, τις βίζα, την βίζα μέχρι τον Απρίλιο. Όμως περιμένουμε η... να τεθεί σε ισχύ και το Omnibus και δεν ξέρω τελικά πότε η συμφωνία αυτή θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ πριν ή μετά την θέση σε ισχύ του Όμνιμπουσο. Θα μπορούσα εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι θα πρέπει οι συμβαλόμενοι να λάβουν υπόψη τους κάθε ε, πληροφορία ε, η οποία μπαίνει στο σύστημα από κάποιον άλλον συμβαλόμενο. Νομίζω δηλαδή ότι αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο θα μπορούσαμε να δουλέψουμε λίγο παραπάνω. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριο Σταβάρες. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. πρόκειται για μια περίπτωση όπου το να δράσουμε άμεσα σημαίνει ότι επηρεάζουμε θετικά την ζωή των πολιτών της ευρωπαϊκής κοινότητας. Και αυτό φαίνεται εδώ και με ένα ιδιαίτερα πρακτικό τρόπο. Το είδαμε εδώ κοντά μας πρόσφατα Είχαμε την περίπτωση ενός φοιτητή από την Αγγόλα, ο οποίος περίμενε να πάρει μια θεώρηση μακράς διαμονής, κάτι το οποίο δεν ήταν εφικτό, γιατί επρόκειτο για έναν πολίτη μιας τρίτης χώρας. Υπήρχε αυτή η έλλειψη δηλαδή δυνατότητας, κινητικότητας για το άτομο αυτό. τώρα πιστεύω ότι η στρατηγική μας είναι καλύτερη, είναι σωστή. Μπορούμε να προχωρήσουμε και να διευκολύνουμε την ζωή πολλών ανθρώπων εγκρίνοντας αυτές τις θεωρήσεις μακράς διαμονής θα μπορούσαμε δηλαδή να διευκολύνουμε την κινητικότητα κάποιων ε, ανθρώπων. Και καμιά φορά τα stickers δεν επιτρέπουν την εισαγωγή βιομετρικών στοιχείων διότι υπάρχει αρνητική θεώρηση αυτής της εισαγωγής. Υπάρχουν άνθρωποι με θεωρήσεις μακράς διαρκείας σε ένα κράτος μέλος δεν θεωρούνται ύποπτα πρόσωπα και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών μελών έτσι ώστε ε, ο κάτοχος μιας τέτοιας θεώρησης μακράς διαρκείας να μην θεωρείται ύποπτος σε ένα άλλο κράτος μέλος έτσι ώστε να ε, μην ε, διακυβεύεται το καθεστώς ενδοκινοτικά. Γι' αυτό δεχόμαστε, δεχόμαστε την ε, πρόταση του εισηγητή και το χρονοδιάγραμμά του. Σας ευχαριστώ τα Ταβάρη. Τελευταία η κυρία Βικοβίτση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Παύλο Κοέλιο. Εξαιρετική δουλειά που έκανε και νομίζω ότι η έκθεση αποτυπώνει με πολύ καλό τρόπο την κοινή επιθυμία μας να εγκρίνουμε το στιμότερο δυνατόν το έγγραφο αυτό. Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην επίλυση των προβλημάτων υπηκών τρίτων χωρών που διαμένουν στα κράτη-μέλη μας ο εισηγητής έθεσε το παράδειγμα ενός υποθετικού φοιτητή στο Βέλγιο. Να θέσει όμως ένα παράδειγμα από τη Λιθουανία. Ένας ε, οδηγός φορτηγού σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορεί να εκτελέσει τη δουλειά του, δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του, γιατί δεν μπορεί να κινηθεί ελεύθερα στην περιοχή Σένιεν. Είναι πολύ καλό το ότι η πρόταση μιλάει για άδειε παραμονής και για θεωρήσεις μακράς διαμονής ως ισότιμης αξίας έγγραφα. Για το πιο σημαντικό εδώ δεν είναι η διάρκεια, η, η χρονική συγκυρία, το πότε μπορεί να μετακινηθεί ο κάτοχος της ε, θεώρησης αυτής εντός της περιοχής Σέγγεν, αλλά η αρχή ότι θα πρέπει το άτομο αυτό να είναι σε θέση να πληρεί και να ικανοποιεί τις ανάγκες του να έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα. Θα ήθελα εκ παραλίλου να πω το εξή. Κοιτώντα τι γίνεται στα κράτη-μέλη, βλέπουμε ότι σε ορισμένε περιπτώσει τα πολιτικά συμφέροντα επηρεάζουν την έκδοση θεωρήσεων τύπου D και C. Θα πρέπει να απλοποιηθεί η διαδικασία για την έκδοση θεωρήσεων. Και επίσης θεωρώ ότι θα πρέπει να συζητήσουμε από το θέμα των ε, δικλείδων ασφαλείας. Γιατί θα πρέπει να διασφαλίσουμε την απλοποίηση αυτή της μετακίνησης των ατόμων αυτών. Είπε πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τηρηθούν οι διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ελπίζω αυτό να το δούμε και στην πράξη. Και θα ήθελα να πω ότι μέχρι 5 Απριλίου του χρόνου θα ήθελα να έχουν επιληθεί όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Ο εισηγητής θα ήθελε να κάνει τα καλλιτικά σχόλια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας και τα σχόλια που έκαναν όλοι οι συνάδελφοι. Επιτρέψτε μου να απαντήσω κυρίως και στην, προς την κυρία Κετάβα Είχε πει. Μας είπε ότι την ανησυχεί το γεγονός ότι θα υπάρχει ε, εισδοχή δεδομένων στο σύστημα Σέγγεν. Να σας υπενθυμίσω ότι η πρότασή μας είναι να μην ενταχθούν ε, αυτοί οι οποίοι ζητάνε θεώρηση ΔΕΛΤΑ στο σύστημα. Απλώς θα πρέπει να εξακριβώσουμε εάν αυτοί οι οποίοι ζητάνε την θεώρηση αυτή συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα Σέγγεν. Δεν θέλουμε να συμπεριλάβουμε περισσότερα ε, δεδομένα, απλώς θέλουμε να εξακριβώσουμε εκ των προτέρων εάν αυτός ο οποίος ζητάει την θεώρηση ΔΕΛΤΑ βρίσκεται ή όχι στο σύστημα. Και αυτό το κάνουμε για λόγους ασφάλειας. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και για να προστατεύσουμε τα άτομα, διότι σήμερα υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν θεώρηση ΔΕΛΤΑ, τα οποία ε, κρατώνται στα σύνορα, διότι έχουν το ίδιο, γιατί κάποιο που έχει το ίδιο όνομα με αυτούς συμπεριλαμβάνεται στο σύστημα Σέγγεν. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Και στην πρόταση μα ζητάμε και το ανάποδο. Δηλαδή, πριν να συμπεριλάβουμε μια κοινοποίηση για την πρόσβαση, την απαγόρευση πρόσβασης στον χώρο Σέγγεν, να εξακριβώνουμε κατά πόσον ο άνθρωπος αυτός έχει ήδη μια θεώρηση Δέλτα. Αυτά τα πράγματα ζητάμε και πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό προστατεύουμε την ελευθερία κυκλοφορίας των πολιτών των τρίτων χωρών αφενός, αλλά και αφετέρου προστατεύουμε και την ασφάλεια του χώρου Σέγγεν. Πρόεδρε, νομίζω ότι θα ήταν καλό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συνεργαστούν μαζί μας αυτές τις δύο εβδομάδες, αυτούς τους δύο μήνες μάλλον. Ε, θα περιμένουμε τις προτάσεις από Πλευρά των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ε, σταυρώσουμε τα χέρια και να μην προσπαθήσουμε να βρούμε μια συμβαστική λύση ανάμεσα στα άλλα δύο θεσμικά όργανα της κοινότητας έτσι ώστε η συμφωνία να επιτεθεί μέσα στα πλαίσια της πρώτης ανάγνωσης. Ε, ελπίζω ότι ότι όλοι οι σκιώδεις εισηγητές και οι εισηγητές των άλλων ε, ε, επιτραπών πιστεύουν ότι θα πρέπει πριν από τις 5 Απριλίου να υπάρξει ε, γνωμοδότηση και θα πρέπει να βιαστούμε. Γι' αυτό ζητώ από το Ευρωπαϊκό, Κοινοβούλιο, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστούν μαζί μας γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε την ασφάλεια αλλά θέλουμε ταυτόχρονα να ενισχύσουμε και την προστασία των δεδομένων και ελπίζουμε ότι η Κομισιό θα μας ε, υποστηρίξει θα υποστηρίξει τις προτάσεις μας και σε αυτόν τον τομέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή, λέει η Πρόεδρος. Υποστεύω ότι το Συμβούλιο και η Κομισιό ε, συμφωνούν να υπάρξει αυτή η διαθεσμική συνεργασία και να συνεργαστούν και με, τον, με τους εισηγητές και τους ισκιώδεις εισηγητές. Από ό,τι κατάλαβα υπάρχει και μια προθεσμία 18 Ιανουαρίου για την υποβολή των τροπολογιών στην έκθεσή σας κύριε Κοέλιο, έτσι ώστε στις 4 Φεβρουαρίου Ιανουαρίου να υπάρξει ψηφοφορία στην Επιτροπή. Σωστά, συμφωνείτε κι εσείς, πολύ ωραία. Εδώ ολοκληρώνεται το σημείο αυτό τη ημερήσία διάταξη. Συνάδελφοι, στις 4 η ώρα, από ό,τι λέει και τα χαρτιά μου εδώ, στις 4 η ώρα θα συναντηθούμε με τον κύριο Άλεξ Τούρκο, που είναι ο πρόεδρος ε, της ομάδας εργασίας του άρθρου 29. Έχουμε επομένω 20 λεπτά στη διάθεσή μας για το επόμενο σημείο. Το λέω αυτό από την αρχή, έτσι ώστε όσοι θέλουν να πάρουν το λόγο να ε, δείξουν μια κάποια πειθαρχία αρχεία και να σεβαστούν τον χρόνο ομιλίε 2 ή έω και 3 λεπτών. σω να μην χρειαστούμε όμω και τόσο πολύ χρόνο. Λοιπόν, το επόμενο σημείο τη ημερήσία διάταξη ε, αφορά την μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Schengen SIS ε, 1 στο SIS 2 στο σύστημα προφοριών Σέγγεν δεύτερης γενιάς. Θα υπάρχουν κάποιες προτάσεις σχετικά με, τα, ε, με τα, εργαλεία, τα νομικά εργαλεία, τα κείμενα τα οποία χρειάζονται για να περάσουμε από το ένα σύστημα στο άλλο. Και αν κατάλαβα καλά, οι προτάσεις αυτές θα αποτελέσουν αντικείμενο συναπόφασης ή όχι. α, θα εκπέσει το κομμάτι που αφορά τον τρίτο πυλώνα. Αλλά τέλος πάντων ας ακούσουμε καταρχάς από τον εισηγητή που είναι ο κύριος Κοέλιο πάλι. Ε, και είναι και η μέρα της Λισαβόνας σήμερα, νομίζω ότι πέφτει πάρα πολύ καλά. Και μετά θα ακούσουμε και τις προτάσεις μου ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω ότι είμαστε πολύ απογοητευμένοι ε, με τις καθυστερήσεις του ΣΥΣ 2. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα στις 22 ε, Οκτωβρίου όπου ε, εκφράζει τις ανησυχίες και τη λύπη του για τις καθυστερήσεις αυτές και μιλά για τα τεχνικά κείμενα τα οποία μας έχουν δοθεί. Καταλαβαίνετε ότι εμπλέκονται πολλοί ε, φορείς και υπάρχουν και νομικές συνέπειες. Το θέμα της μετανάστευσης είναι πολυσχηδές. Θα πρέπει να ξέρουμε κατά πόσο υπάρχει μία ημερομηνία αναστολής. Δηλαδή, η Επιτροπή μας προτείνει μία λευκή επιταγή διαβίου. Δεν υπάρχει προθεσμία, καταληκτική ημερομηνία, ε, η οποία θα πρέπει να εισαχθεί. Εμείς δεν δίνουμε λευκές επιταγές, θέλουμε μια διαδικασία με σαφές χρονοδιάγραμμα. Επίσης, η μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να εξεταστεί από το Κοινοβούλιο. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τη νομική βάση του ΣΥΣ από δημοσιονομικής πλευράς, γι' αυτό θα θέλαμε να συνοδεύσουμε αυτή την αρχή και διαδικασία με μεγάλη αυστηρότητα. Γι' αυτό, πριν από τη μετάβαση προς ένα νέο σύστημα, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται επαρκώς και να γνωμοδοτεί θετικά. Από την άλλη πλευρά, Κανένας μας δεν έχει εγγυήσεις ότι το ΣΥΣ 2 θα ανακύψει όπως προβλέπεται. Πρόκειται για κείμενα που θα αξιολογηθούν. Άρα, ίσως θα πρέπει να αρκεστούμε σε μια τεχνική λύση που είναι διαφορετική από το ΣΥΣ2. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι εάν, εάν γίνει κάτι τέτοιο, αν έχουμε μια διαφορετική δηλαδή τεχνική λύση, όλες οι νομικές διατάξεις θα πρέπει να υφίστανται σε αυτή τη νέα τεχνική λύση. Δεν θα πρέπει δηλαδή να προβούμε σε ένα βραχικύκλωμα, σε μια ε, βραχικύκλωση του ΣΥΣ 1. Υπάρχει και το Global Program Management Board όπου ε, έχουμε δύο οκτώ τεχνικούς από τα κράτη-μέλη και δύο από την Κομισιό. Λυπάμαι διότι το Global Management Board δεν αποφασίστηκε εξ αρχής. Έτσι θα είχαμε αποφύγει μερικά προσκόμματα εάν είχαμε ζητήσει την αρρωγή των εμπειρογνωμόνων από τα κράτη-μέλη χωρίς να υπάρχουν αντιπαλότητες, ανεπιθύμητες αντιπαλότητες. Εν συμπεράσματι, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι εάν το προσχέδιο ΣΥΣ 2 δεν προωθηθεί, εάν υπάρχει αρνητική έκβαση δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται να καλέσει το ελεγκτικό συνέδριο έτσι ώστε να εξεταστεί η διαχείριση του σχεδίου ΣΥΣ 2, ιδιαίτερα ως προς τις ε, δημοσιονομικές επιπτώσεις. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω σε σχέση με τις θεωρήσεις μακράς διαρκείας, η κατάσταση είναι η ίδια και τέλος μόλις πληροφορήθηκα ότι στη συνάντηση του Συμβουλίου ΖΑΗ αναβλήθηκε για άλλη μια φορά το συνολικό κείμενο του Milestone 1 που θα αποφασιστεί στα τέλη Ιανουαρίου. Επίσης, το Συμβούλιο τόνισε ότι αν δεν εγκριθούν τότε αυτά τα κείμενα Δηλαδή, αν ε, δεν ε, καταλήξουμε στα τέλη Ιανουαρίου, το Συμβούλιο θα συμπεράνει ότι το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Θα ήθελα η Επιτροπή και το Συμβούλιο να μας δώσουν νέες πληροφορίες σε σχέση με το χτεσινό Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κοέλιο. Θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν τον κύριο ή την κυρία Τιντοράτσι να απαντήσουν στα σχόλια του κυρίου Κοέλιο. Ο κύριος Τιντοράτσι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισήγητη για την εκτενή παρουσίαση και συμφωνώ με τις πολλές επιφυλάξεις που προανακοίνωσε. Ίσως πριν μπω στην παρουσίαση καθεαυτή, γιατί ξέρω ότι πιεζόμαστε από το χρόνο. Νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να σας ε, μιλήσω για τη χθεσινή συνάντηση και να σας δώσω και ορισμένες πληροφορίες που δεν ε, γνώριζε ο εισήγητης. Και να σας πω ότι την τελευταία φορά τη εισήγησης του κυρίου Μπαρό ε, στην Ολομέλεια μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς τις συμβάσεις ε, που θα έπρεπε να συναφθούν μέχρι το τέλος του έτους, μέχρι το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας φτάσαμε σε μια συμφωνία ε, με τους συμβασιούχους να συνεχίσουν με τις δοκιμές και εάν δεν είναι επιτυχής τότε θα πρέπει να κινηθούμε στο εναλλακτικό σενάριο σε σχέση με τους ε, θεσμικούς μηχανισμούς του Συμβουλίου που αποφασίστηκαν φέτος τον Ιουνίου. Οι δοκιμές αναβλήθηκαν για τις 29 Ιανουαρίου και το χτεσινό Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων θεώρησε ότι αν δεν τηρηθεί αυτή η προθεσμία, τότε το Συμβούλιο μέσα σε δύο μήνες θα αποφασίσει για το πώς θα εκκινηθεί το σύστημα. Ως προς τα μέσα που διαθέτουμε για τη μετανάστευση. Όπως είπε ο κύριος ε, Κοέλιο, μέχρι τα τέλη Ιουνίου λήγουν τα μέσα μετανάστευσης και το Συμβούλιο του Ιουνίου κάλεσε την Επιτροπή να θεσμοθετήσει το Global Project Management Board, που ήταν μια άτυπη ομάδα η οποία συστάθηκε από το Συμβούλιο στις αρχές του έτους. Και συμφωνώ με τον κύριο Κοέλιο ότι δηλαδή η εμπειρία μας ήταν πολύ θετική και έχουμε βελτιώσει την ε, συνεργατική προσέγγιση κατά τη διαχείριση του σχεδίου αυτού. Και έτσι η θεσμοθέτηση ήταν ε, το φυσικό απότοκο της ε, όλης κατάστασης. Αυτό αποφασίστηκε από το Συμβούλιο του Ιουνίου και η νομική ευελιξία θα πρέπει να εισαχθεί στη νομική βάση για την αλλαγή στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης εάν αποτύχουν οι δοκιμές. Άρα αυτή είναι η εντολή μας και τροποποιήσαμε τα μέσα μετανάστευσης, Migration Instruments. Θα αλλάξουμε το τρέχον κείμενο και θα έχουμε ένα άρθρο που περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που έχουμε προβλέψει θα ήθελα να δω μία προς μία. Ως προς τη νομική ευελιξία στην οποία προαναφέρθηκε το αναλλακτικό σχέδιο, η προσέγγιση μας σχετίζεται με αυτά που προείπε ο κύριος Κοέλιο και αυτό το επικύρωσε και το Συμβούλιο του Ινιού και η νομική μας υπηρεσία. Δηλαδή, ε, θα πρέπει να έχουμε μια λειτουργική προσέγγιση όταν προετοιμάζουμε τη νομική εργασία για αυτή την ε, μετάβαση και ε, δυνάμει αυτή της ε, λειτουργικότητας, των κανόμενων, κανόνων λειτουργικότητας, θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία για οποιασδήποτε άλλες τεχνικές λύσεις, έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτές τις επιμέρους λειτουργικότητες, τη στιγμή που η τεχνική λύση δεν είναι εφικτή. Επομένως, με αυτή την ε, προσέγγιση κατά νου εξετάσαμε τα ε, κείμενα που αφορούν την ε, μετάβαση και προσπαθήσαμε να εξαφανίσουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία εμποδίζουν την νομική δυνατότητα να λειτουργήσει σωστά και να γίνει η μετάβαση σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις. Ναι, μεν είναι δύσκολο αυτό καταρχάς, αλλά προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη μας αυτό το οποίο ονομάζουμε converter που είναι ε, αυτός, αυτό το οποίο επιτρέπει να γίνει η μετάβαση αυτή και να ξεπεράσουμε τις ε, τεχνικές δυσκολίες. Δηλαδή μπορέσαμε να εισάγουμε την απαραίτητη ευελιξία. Τώρα ε, για το GBMB είδαμε τι δουλειά έχει κάνει η ομάδα μέχρι τώρα και εισάγαμε στο κείμενο τις απαραίτητες διατάξεις ε, έτσι ώστε να, γίνει, να, να γίνει εφικτή η μετάβαση. Τώρα, καταλαβαίνω τις ανησυχίες του κυρίου Κοέλιου όσον αφορά την ημερομηνία. Εμείς θεωρήσαμε ότι έτσι όπως έχουν τα πράγματα τώρα δεν ξέρουμε ποιος είναι ο, ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε διότι τα πάντα εξαρτώνται από την ε, επιτυχία της δοκιμής που θα γίνει τέλος ε, Ιανουαρίου. Όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα τώρα γιατί δεν έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία στη διάθεσή μα. Γι' αυτό είπαμε να υπάρχει μια ανοιχτή ημερομηνία και τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα στο Συμβούλιο ανάλογα με την λύση που θα επιλεγεί τελικά να αποφασίσουμε ποια θα είναι η οριστική ημερομηνία. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Ένσο, ζητήσατε το λόγο, αλλά να είστε λίγο σύντομος, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Είμαι σκιώδης και εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι η εργασία του κυρίου Κοέλιου ήταν ε, εξαιρετική. Θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να μας δώσει μια συγκεκριμένη ημερομηνία έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το project θα τεθεί σε εφαρμογή. Θα γίνουν οι ε, δοκιμές, αλλά υπάρχουν πολλοί υποθετικοί λόγοι, δηλαδή αν επιτύχουν οι δοκιμές, αν προωθηθεί το κείμενο, αν, αν. Δηλαδή αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχουν σαφείς όροι για να τεθεί σε εφαρμογή αυτό το πλαίσιο. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι καταβλήθηκαν και, πολλές, και πολλά χρήματα. Υπήρξαν πολλές δαπάνες και η Επιτροπή θα πρέπει να μας υποβάλει μια πρόταση σε σχέση με τα συγκεκριμένα ζητήματα ως προς την προστασία προσωπικών δεδομένων των πολιτών που είναι ύψης της σημασίας. Θα συνεργαστούμε με τον κύριο Κοέλιο και νομίζω ότι θα καταφέρουμε κάτι το καλό. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελε κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Ε, αν όχι, ξαναδίνω το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι μπορώ να προσθέσω τίποτα στη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τις άλλες πολιτικές ομάδες για την υποστήριξή τους. Νομίζω ότι η θέση του Κοινοβουλίου είναι σαφέστατη επί του θέματος. Χρειαζόμαστε τη δεύτερη γενιά ε, του συστήματος πληροφοριών Σέγγεν. Πρέπει να ενισχύσουμε την, το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών μας και είμαστε απογοητευμένοι με τις καθυστερήσεις ε, που παρουσιάζει όλη αυτή η διαδικασία. Κατανοούμε την ανάγκη ότι χρειάζονται τα απαραίτητα κείμενα για να γίνει αυτή η μετάβαση. Ε, δεν μας αρέσουν κάποιες από τις διατάξεις που προτείνει η Κομισιό. Ε, κάναμε τις απαραίτητες τροπολογίες, οι προτάσεις για τροπολογίες και ελπίζουμε ότι θα έχουμε την δυνατότητα να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία αφού ακούσουμε και τις συνεισφορές των Εθνικών Κοινοβουλίων. Διότι και εδώ, σε αυτόν τον τομέα, περιμένουμε την τις ε, προτάσεις ε, των κοινοβουλίων. Για 8 εβδομάδες πρέπει να περιμένουμε. Ε, πάντως πιστεύουμε ότι η προστασία των δεδομένων είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά θέματα με τα οποία ασχολεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ λέει η Πρόεδρος. Στο επόμενο, το επόμενο σημείο της, της ημερήσιας διαταξής μας είναι το σημείο 10, συνάντηση με τον κύριο Άλεξ Τούρκο, πρόεδρο της ομάδας εργασίας του άρθρου 29, ο οποίος είναι εδώ. Yes, Mr. Mr. Turk, very welcome to our, to our committee. Σας καλωσορίζω κύριε Τούρκο στην Επιτροπή μας και μια τέτοια σημαδιακή ημέρα που είναι η θέση σε ισχύ, σε λειτουργία της συνθήκης της Λισαβόνας, που θα, μια συνθήκη που αλλάζει το όλο καθεστώς της προστασίας των δεδομένων. Ε, γι' αυτό θα θέλαμε να ακούσουμε τις απόψεις σας για αυτό το νέο καθεστώς όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Έχει το λόγο κύριε Τούρκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ε, καλωσορίζετε εδώ στην, ε, στην Επιτροπή σας για να προχωρήσουμε σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Να πω ευθύς εξ αρχής ε, ότι θα εκφράσω τις προσωπικές μου απόψεις λίγο πολύ, διότι ναι μεν είμαι ακόμα πρόεδρος της ομάδας εργασίας, αλλά για λίγες μέρες αυτής θα είμαι πρόεδρος της ομάδας εργασίας για το άρθρο 29. Και ο λόγος για τον οποίο δεν θα παραμείνω πρόεδρος ε, θα ε, είναι ε, το αντικείμενο της ομιλίας μου. Αποφάσισα να μην υποβάλλω ξανά υποψηφιότητα και αποφάσισα επίσης να διευκολύνω την ε, ζωή του διαδόχου μου λέγοντάς σας τι δεν πάει καλά. Αλλά αυτά είναι προσωπικές μου απόψεις. Ε, αυτές θα εκφράσω τώρα και δεν θα μιλήσω εξ ονόματος όλης της ομάδας εργασίας γιατί δεν το έχουμε συζητήσει. Είναι ένα είδος κληρονομιάς διαθήκης που αφήνω. Ε, να σας πω τι αισθάνομαι έτσι ενστικτοδός σήμερα. Γιατί 17 χρόνια ασχολούμαι με το θέμα των προσωπικών δεδομένων και σαν πρόεδρος αρμόδιας επιτροπής στο Παρίσι και σαν ε, βουλευτής αλλά και σαν πρόεδρος ομάδας εργασίας του άρθρου 29 εδώ και δύο χρόνια. Να σας πω πόσο μπορεί να προχωρήσει η λειτουργία της ομάδας αυτής για να διευκολύνουμε και τη ζωή μας. Η πρώτη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι ότι ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα ότι το θέμα Τη προστασία ε, της των προσωπικών δεδομένων είναι, είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, περισσότερο από ό,τι ε, φανταζόμαστε εμείς, διότι είναι, αποτελεί ακριβώς την καρδιά της δημοκρατίας. Έχουμε την, ε, την το, την αίσθηση ότι η δημοκρατία σημαίνει ότι η, το, το, το καθεστώς πρέπει να είναι διάφανο. Η κυβέρνηση πρέπει να ε, δρά με έναν διάφανο τρόπο. Για να μπορεί να γίνει αυτό υποτίθεται ότι η κυβέρνηση πρέπει να έχει πρόσβαση στις διάφορα αρχεία. Ο στόχος, ο στόχος των ε, δικών μας ε, τέτοιων νομικών εργαλείων είναι να διαφυλάξουμε την προσωπική ζωή των πολιτών. Τώρα, η η διαφάνεια της κυβέρνησης δεν εξαρτάται από μας, εξαρτάται από την αστυνομία και εκείνοι ασχολούνται περισσότερα με τα θέματα των αστυνομικών φακέλων κτλ. Εξού και εγώ θα ασχοληθώ μόνο με αυτά τα οποία απασχολούν περισσότερο την ομάδα ε, εργασίας του άρθρου 29. Αυτό το οποίο με ανησυχεί περισσότερο σήμερα στο σύνολο των χωρών και όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτό το οποίο ονομάζω διπλή ίχνη λασιμότητα, διπλά ίχνη. Ούτως ή άλλως μπαίνουμε σε αυτή την ψηφιακή κοινωνία κοινωνία όπου το σύνολο των πολιτών μας και όχι μόνο στην Ευρώπη θα πρέπει συστηματικά είτε το θέλουν είτε όχι και καμιά φορά το θέλουν, καμιά φορά δεν το θέλουν όμως μερικές φορές το ξέρουν, μερικές φορές δεν το ξέρουν ε, λοιπόν καλούνται να να αποτελούν αντικείμενα παρακολούθησης από μακριά ενδεχόμενα. Εξού και υπάρχει αυτή η, η, χνηλασιμότητα, αυτή η παρακολούθηση, αυτή, ε, ε, αυτό γίνεται μέσα από δίκτυα. Χτες κάναμε μια κρόαση για ε, κάποια κοινωνικά δίκτυα, τα social networks ε, και το πρόβλημα ήταν πώς ένα άτομο το οποίο είναι 19-20 χρόνων που λέει κάποια πράγματα που εκφράζεται μέσα στο δίκτυο μετά από λίγα χρόνια να ε, βρει την ελευθερία του. Να μην τον παρακολουθούν εσαΐ για αυτά τα οποία είπε ή έκανε κάποια δεδομένη στιγμή. Και αυτή, αυτό που θίγεται εδώ αυτή τη στιγμή είναι η έκφραση ελευθερίας, η δυνατότητα που έχεις να οριμάσεις, να αναπτυχθείς, να εξελιχθείς. Εδώ πιστεύω ότι χάνουμε αυτή την δυνατότητα που έχουμε της ελευθερίας έκφρασης. Ένα αυτό. Δεύτερον, όλα αυτά τα ε, οι, μηχανές ε, έρευνα ε, εκεί μπορούμε να, βρούμε στοιχεία τα οποία ελέγχουν, αν θέλετε, τις, ε, τις ε, δραστηριότητές μας. Από την άλλη πλευρά έχουμε να κάνουμε με την βίντεο επίβλεψη, με την, με την παρακολούθηση των, της κίνησης των ανθρώπων και των αγαθών τα βιομετρικά στοιχεία. Εδώ το άτομο μπορεί να αποτελεί αντικείμενο παρακολούθησης, να το, να το ακούνε, να το εντοπίζουν, να εντοπίζουν τις, ε, τις κινήσεις του γίνεται μια φυσική δηλαδή παρακολούθηση. Επομένως η προσωπική ζωή σιγά σιγά εξαφανίζεται. Η προσωπική ζωή και είναι μια, δεν είναι μια κοινωνική, είναι μια μάλλον κοινωνική λειτουργία. Μας επιτρέπει να ζούμε μέσα στα πλαίσια μιας κοινωνίας σεβόμενοι η μεν τους δε. Εάν όμως όλοι παρακολουθούν τις προσωπικές ε, σεξουαλικές συναισθηματικές ε, εκφράσεις μας και εκδηλώσεις μας, τι γίνεται με την ελευθερία μας, πού βρίσκεται αυτή η προσωπική ελευθερία σε καθημερινή βάση. Το πρόβλημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων δεν είναι τεχνικό θέμα, αποτελεί ένα θέμα που είναι η καρδιά της ε, κοινωνίας μας, διότι είναι ένας μηχανισμός ο οποίος μας επιτρέπει να ζούμε ευτυχισμένοι και οι μεν και οι δε σε μια ψηφιακή κοινωνία. Και αυτό είναι, πάρα, είναι ελάχιστο γνωστό σήμερα. Και είμαι εδώ για να σας πω ότι κάθε μέρα που περνάει ενδυναμώνει και ενισχύει την αγωνία μου. Διότι πραγματικά έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε γίνει κατανοητοί πάνω σε αυτό το θέμα. Και μας παρακολουθούν παντού. Ε, μας αντιμετωπίζουν σαν ε, κάποια άτομα τα οποία είναι λίγο περίεργα, τα οποία ε, έχουν μια αιμονή με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όμως εμείς πιστεύουμε ότι αυτά είναι ε, τα στοιχεία που θα μας επιτρέψουν κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουμε γυρίζοντας προς τα πίσω ότι έχει αλλάξει τελείω η κοινωνία μας και κάνω και μια, ένα παραλληλισμό ανάμεσα στην προστασία του πλανήτη και την προστασία του, δικού μας πλανήτη, του, του, του, του, προσωπικού μας πλανήτη αν θέλετε, της, της ζωής μας. Διότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πώς ζούμε, ποιο είναι το περιβάλλον. Ε, το, και αυτό το περιβάλλον έχει αλλάξει ε, και δεν μπορούμε εμείς να το ανασαστήσουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να εμπνευστούμε από όλη την, ε, την προβληματική του περιβάλλοντος και του περιβάλλοντο του πλανήτη μας δηλαδή και να διασφαλίσουμε και τον δικό μας πλανήτη, τη δική μας ζωή. Υπάρχουν κάποιες απαντήσεις βέβαια που μπορούμε να, βρούμε. παραδείγματο χάρη σε τεχνολογικό επίπεδο. Θα βρούμε τεχνολογικά, τεχνολογικές απαντήσεις. Το δεύτερο είναι οι, οι ενέργειες που αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, σε νομικό επίπεδο, ε, στα διάφορα κράτη-μέλη της κοινότητας. Επίσης, ε, θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο κοινοβουλευτικός αντίκτυπος ε, των ε, των ενεργειών που κάνουν τα κοινοβούλια σε εθνικό επίπεδο. Γιατί τα κοινοβούλια δεν κάνουν καμία μελέτη αντικτύπου των διαφόρων μέτρων που υιοθετούνται για τα αρχεία κτλ. Επίσης, θα πρέπει αναγκαστικά να ενημερώσουμε και να εκπαιδεύσουμε τους νέους έτσι ώστε να μπορούν οι νέοι μας γνωρίζοντας ε, όλες τις λεπτομέρειες να κάνουν τις σωστές επιλογές ε, της τεχνολογίας. Επίσης ε, πρέπει να γίνει πάρα πολύ δουλειά και αυτό το κάνανε και κάποιοι αρχές μας στη Μαδρίτη εδώ και μερικές εβδομάδες γιατί 80 αντιπροσωπείε συμφώνησαν πάνω σε ένα σώμα βασικών αρχών. Αυτή είναι, αυτό είναι ένα πρώτο βήμα, ουσιαστικό βήμα, το οποίο ε, σημαίνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Πρόκειται όμως για ένα πρώτο βήμα. Μετά ακολουθεί ένα άλλο βήμα, ένα άλλο στάδιο πολύ πιο δύσκολο, το οποίο θα απαιτήσει ε, και μία πολιτική θέληση μεγαλύτερη, που είναι η αναγνώριση της δεσμευτικής νομικής ε, αξίας αυτών των διατάξεων. Αυτό όμως χρειάζεται κάποια χρόνια για να γίνει. Εν τω μεταξύ όμως η τεχνολογία προχωράει και εφαρμόζεται. Και επίσης υπάρχει και ο ρόλος, τον οποίο παίζουν συγγνώμη, ε, κάποια θεσμικά όργανα, παραδείγματο χάρη αυτό της ε, ομάδας εργασίας ε, του άρθρου 29, του οποίου, της οποίας προεδρεύω. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναλάβουμε τρει αποστολέ. Η πρώτη αποστολή μα τη γνωρίζετε, θα πρέπει να απαντήσουμε στα αιτήματα τα οποία μα υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσπαθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αυτό νομίζω ότι το κάνουμε μέσα από μια πολύ καλή δουλειά, πολύ υψηλή ποιότητα δουλειά, να γνωμοδοτήσουμε, να δώσουμε τι τις συμβουλέ μας κτλ. Δεύτερον, να έχουμε μία, έναν ρόλο ιδίε πρωτοβουλίες. Θα πρέπει δηλαδή να αναλάβουμε πρωτοβουλίες από μόνοι μα. Όταν διαπιστώνουμε ας πούμε ότι το σύνολο των οργανώσεων ίσω σε όλο τον κόσμο ε, εφαρμόζει κάποιες προδιαγραφές που στηρίζονται απλώς και μόνο στον περιορισμό ε, την, ε, του ΟΠΕΚ ή ε, ε, του ΟΣΑ ας πούμε ε, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς λέμε και τι ακριβώς κάνουμε. Τρίτον όμως, θα πρέπει η ομάδα μας, αλλά δεν έχουμε το χρόνο για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να παίξουμε και έναν ρόλο σε σχέση με τα ίδια τα κράτη και τους ίδιους αρχές και τις αρχές ελέγχου των κρατών γιατί δεν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ενδεχόμενα να υπάρχουν και κάποιες ανισότητες ε, γιατί κάποιες αρχές ελέγχου ασκούν πραγματικές, ε, ε, πραγματικό έλεγχο άλλες χώρες αναπτύσσουν απλώς εκπαιδευτικές πολιτικές ε, όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα αλλά το θέμα είναι μήπως θα πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω και όλα τα κράτη να προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το σύνολο των εργαλείων που έχουν στη διάθεσή τους και εδώ η ομάδα του Ιάρθρου 29 έχει να παίξει έναν σημαντικό ρόλο ένα ρόλο όμως ο οποίος δεν καθορίζεται από τα κείμενα αυτό το οποίο με ανησυχεί πάρα πολύ είναι η απουσία μέσων και αυτό είναι κραυγαλαίο. Τώρα, το λέω τώρα που εγκαταλείπω ε, την Προεδρία και την εγκαταλείπω γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Και αυτό, αυτή είναι μια ευθύνη την οποία αναλαμβάνω. Και θεωρώ ότι ε, βοηθάω αυτή τη στιγμή τον ε, διάδοχό μου το, η Επιτροπή του άρθρου 29 μπορούν να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα και για άλλα θέματα, για το SWIFT ή οτιδήποτε. Για να τα κάνει όλα αυτά όμως χρειάζεται κάποιο προπολογισμό. Όμως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα κονδύλι. Γι' αυτό θα ήθελα να ξέρω πώς μια οργάνωση μια τέτοια φύσης θα μπορούσε να αναπτύξει ενέργειες και δραστηριότητες, να κάνει, να κάνει ακροάσεις, να δίνει τις ε, ε, γνωμοδοτήσεις της, να οργανώνει κάποιες ομάδες εργασίες, να επισκέπτεται ε, κάποιους χώρους χωρίς να έχει κανένα προπολογισμό. Πολλές φορές ζητάμε μέσα για να κάνουμε κάποιες εμπειρογνωμοσύνες, αυτό βέβαια δεν συμβαίνει συχνά, αλλά πώς μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας εάν δεν έχουμε το ελάχιστον ε, της αυτονομίας. Παραδείγματος χάρη σήμερα έκανα έναν υπολογισμό στην η, Εθνική Επιτροπή τη Γαλλία ε, και ελπίζω να μην υπάρχουν πολλοί Γάλλοι μέσα στην αίθουσα, αλλά εφόσον δεν έχουμε προϋπολογισμό για τους Γάλλους και τα δύο χρόνια της Προεδρίας μου μας κόστησε η, η Επιτροπή αυτή του άρθρου 29 150.000 ευρώ. Επομένως διορωτώ με, μπορεί κάποιος εκπρόσωπος μιας μικρής χώρας να αναλάβει την Προεδρία της, ε, του άρθρου 29. Όχι βέβαια. Και επομένως, αν δεν κάνουμε κάτι, πρόεδρος της ε, ομάδας αυτής θα είναι κάποιος που προέρχεται από μια μεγάλη χώρα, που να μπορεί να καλύψει τα έξοδα. Και αυτό το θεωρώ απαράδεκτο και πριν να ολοκληρώσω για να ακούσω τις ερωτήσεις σας, θα ήθελα να σας πω ότι πάρα πολύ συχνά ανησυχούμε για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, έγινε ένας, ζητήθηκε ένας έλεγχος ε, της Επιτροπής, της ομάδας μας και απήντησα στα στα ερωτήματα τα οποία ετέθηκαν μέσα στα πλαίσια του ελέγχου. Όμως πρέπει να σας πω ότι μου, έκαναν, μου, έκανε εντύπωση, μου ερωτήσεις διότι προσπαθούς, προσπάθησα να δω τι πάει καλά ή τι δεν πάει καλά. Θα έπρεπε για να δούμε τι δεν πάει καλά ε, θα ήθελα οι ερωτήσεις αυτές να αφορούν την ε, το κατά πόσον θα πρέπει να συνεχίσει η, ε, η ζωή της ομάδας αυτής. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αν θέλουμε να διατηρήσουμε στη ζωή αυτή την ε, ομάδα θα πρέπει να έχει στην διάθεσή της τα απαραίτητα κονδύλια. Πάντως ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξετάσει και την ε, δυνατότητα να δημιουργηθεί μία ομάδα εμπειρογνωμόνων που, θα εκπροσωπούνταν ε, οι, Αμερικανοί και εμείς και κάναμε πραγματικά μια, ένα διάβημα εναντίον της Κομισιόν ε, διότι εμείς κάναμε μια γνωμοδότηση η οποία είναι πάρα πολύ εμπεριστατωμένη και θα δημοσιευθεί μέσα στα πλαίσια της διαβούλευσης που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά τέλος πάντων αυτό το οποίο σημειώνω είναι ότι έπρεπε να αντιδράσουμε εντονότατα γιατί οι Αμερικανοί οι Αμερικανοί ενδεχόμενα να πρέπει να αλλάξουν την νομοθεσία τους. Αλλά ποιοι θα είναι, ποια θα αυτή η ομάδα η οποία θα εξετάσει τις ανάγκες αυτές. Αποτελείται από ποια θα, ποια θα είναι η σύνθεση σε Αμερικανών και Ευρωπαίων στην, στην Επιτροπή αυτή. Επαναλαμβάνω, για να τελειώσω, ότι η εντυπωσία εντυπώσεις αυτές τις οποίες εγώ εξέφρασα είναι προσωπικές εντυπώσεις. Δεν μπορώ να φραστώ εξ ονόματος ε, της ε, ομάδας εργασίας του άρθρου 29. Ε, εύχομαι κάθε τύχη στον διάδοχό μου, θέλω να τον βοηθήσω γιατί οι φάκελοι και τα θέματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πάρα πολύ δύσκολα. Σας ευχαριστώ. Ούτως ή άλλως Είμαστε εδώ για να σας ε, υποστηρίξουμε ηθικά τουλάχιστον. Ε, μιλήσατε με ιδιαίτερο πάθος και αυτές είναι οι τελευταίες μέρες της Προεδρίας σας. Ε, επομένως φεύγετε δημιουργώντας ένα μεγάλο μπαντ Νομίζω ότι η έκκλησή σας ακούστηκε από τα μέλη της Επιτροπής μας, γιατί πολλά από αυτά τα οποία είπατε εσείς ε, είναι και ανησυχίες τις οποίες έχουμε εκφράσει τα τελευταία χρόνια. Και ελπίζουμε ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, τώρα να έχουμε στη διάθεσή μας ε, τα μέσα που θα επιτρέψουν στη φωνή μας να ακουστεί. Τώρα βέβαια τα πάντα εξαρτώνται και από το Κοινοβούλιο. Έχουμε την αντοχή Έχουμε και την ε, δυνατότητα να αντισταθούμε στις πιέσεις ε, που μπορεί να περάσουν από το Συμβούλιο ή από την Κομισιό. Λοιπόν, ποιος συνάδελφος ζητάει το λόγο. Στο Ενωμένο Βασίλειο έχουν, ε, έχει αλλάξει η νομοθεσία και επιμένουμε προκειμένου να φυλάσσονται όλες οι επικοινωνίες μέσω email για δύο χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για πολιτικές επαφές που μπορεί να έχουν οι πολίτες και πολύ. Ναι, μισό λεπτό λέει η Πρόεδρος, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με, την, ε, με τα ακουστικά και τη διερμηνία. Αν θα θέλετε να ξεκινήσετε από την αρχή. Στο Ηνωμένο Βασίλειο λοιπόν τροποποιήθηκε πρόσφατα νομοθεσία και επιμένει προκειμένου όλες οι επαφές ε, ε, email και οι επισκέψεις στους σελίδες να κρατούνται για δύο χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος μπορεί να ελέγχει πολιτικές και λοιπές επαφές των πολιτών και ιδιαίτερα οι κρατικοί υπάλληλοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν επαφές τις οποίες αποδοκιμάζει το κράτος μπορεί να έχουν την αίσθηση ότι ενδεχομένως να ε, πληχθούν και οι καριέρες τους, οι σταδιοδρομίες τους και η δημοκρατία και η ελευθερία του συνέχερστε όχι μόνο στην ε, σωματική της ε, μορφή αλλά και σε όλες τις μορφές είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει λοιπόν τα δημοκρατικά δικαιώματα να μην αποτελούν κενό γράμμα. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω ποια είναι η δική σας άποψη από αυτού. Ευχαριστώ, η Σάρα Λάτφορτ. Και εγώ συμφωνώ μαζί σας πρόεδρε ότι η παρουσίαση την οποία μόλις ακούσαμε και θα πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρά τις δηλώσεις του κυρίου Τούρκ γιατί άλλωστε παρατείται λόγω της έλλειψης ε, συνεργατών σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό και θα πρέπει να πω και να ομολογήσω ότι σε κάποιο βαθμό δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες γιατί υποθέτω ότι δεν υπάρχει χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το, την Επιτροπή του άρθρου 29. Δεν το ήξερα αυτό. Θεωρούσα ότι θα υπήρχε τέτοια υποστήριξη, αλλά φαίνεται ότι το θέμα είναι να συλλέξουμε χρήματα από τα κράτη-μέλη, από τη Γαλλία, οι γαλλικές αρχές σε συγκεκριμένη περίπτωση. Είχαν τα χρήματα να υποστηρίξουν την εργασία του κυρίου Τούρκ κατά την προεδρία του. Αυτή η πρόκληση σαφώς είναι κάτι το παράδεκτο. Δεν ξέρω ποιες είναι οι νομικές ε, προαπαιτήσεις για την χρηματοδοτική ενίσχυση από τον κοινωτικό προϋπολογισμό, αλλά σίγουρα θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Και νομίζω ότι η αναλογία με την αλλαγή του κλίματος είναι πολύ σωστή. Γιατί, αν δεν το ελέγξουμε, δεν μπορούμε να το ανατρέψουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ή μη αδύνατο. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να περιορίσουμε τη ζημιά. Και συμφωνώ απόλυτα ότι βρισκόμαστε πραγματικά σε ένα πολύ κρίσιμο, σε μια πολύ κρίσιμη χρονική συγκυρία σε ό,τι αφορά την, τα προσωπικά δεδομένα. Και αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι η προθυμία των νέων να θέσουν σε κίνδυνο τα προσωπικά τους δεδομένα, δημοσιεύοντάς τα σε ιστοσελίδες. Κινδυνεύουμε δηλαδή να χάσουμε αυτή την πολιτισμική σύνδεση με τα ιδιωτικά αυτά δεδομένα, το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό σε ό,τι αφορά τους πόρους για τις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων ατομικά, ξεχωριστά, θεωρώ ότι η Επιτροπή απείλησε με διαδικασίες επί παραβάση κατά του Ηνωμένου Βασιλείου και του σχετικού αρμοδίου και αυτό έχει οδηγήσει σε αποτελέσματα. Αυξήθηκαν οι σχετικές αρμοδιότητες. Δεν ξέρω τελικά σε ποιο βαθμό προχώρησαν αυτές οι διαδικασίες, αλλά σίγουρα θα υπάρξουν και αποτελέσματα σε άλλες ε, χώρες. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται και έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα με πολλά κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά υποχρεώσεις που δεν έχουν εκπληρωθεί, αλλά πρόκειται για ένα από τα πολύ σημαντικά μέτωπα και αυτό. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση όπου είναι απαραίτητο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από πλευρά τη Επιτροπή μα, αλλά και πάλι ίσω υπάρχουν περιορισμοί, επαναλαμβάνω, χρηματοδοτικοί. Από πλευρά ε, κινητικού προπολογισμού. Ίσως πρόκειται για διακυβερνητική υπηρεσία. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να δούμε τι γίνεται. Ευχαριστώ, Σάρα, λέει η πρόεδρο Πρωτού δώσω το λόγο στην κυρία Ένστ. Νομίζω ότι χρήσιμο θα ήταν να διευκρινιστεί το θέμα αυτό, γιατί αν σωστά κατάλαβα, η ομάδα εργασίας διευκολύνεται από τον... Ε, μάλλον χρησιμοποιεί τον προϋπολογισμό της Επιτροπής. Άρα η Επιτροπή, στην Επιτροπή εναπόκειται να λάβει την απόφαση να διευκολύνει τις εργασίες της Επιτροπής άρθρο 29. Αυτό λοιπόν θα ήθελα να, να μου το επιβεβαιώσετε. Επίσης θα ήθελα να διευκρινίσετε. Είπατε αν ο πρόεδρος της Επιτροπής άρθρο 29 προέρχεται από μια χώρα, η χώρα αυτή θα καλύψει το κόστος της προεδρίας της ομάδας εργασίας, εκτός δηλαδή του προϋπολογισμού της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ομάδα G29 έχει να κάνει, η ομάδα του άρθρου 29 συγγνώμη, είναι κάπως μια ιδιαίτερη ομάδα, ιδιόρυθμη θα έλεγα σε σχέση με τις άλλες ομάδες εργασίες και ε, είναι εκεί για να βοηθήσει την Κομισιόν στις ενέργειές της. Επομένως, εάν πρέπει να έχει κάποια κονδύλια, τα κονδύλια αυτά πρέπει να προέλθουν από την Κομισιόν. Τώρα, για την Προεδρία, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι έπρεπε να οργανώσουμε πούμε, κάποιες ομάδες, ε, κάποιες συνεδριάσεις εργασίας ε, για προβλήματα που αφορούν ε, ας πούμε, τους κανόνες λειτουργίας των εταιριών, που είναι θέματα που είναι πολύ σημαντικά για μας και που περιμένουν από εμά να, να γνωμοδοτήσουμε οι διάφορες εταιρείε. Αυτές είναι συνεδριάσεις που εμείς οργανώνουμε. Εγώ τις είχα οργανώσει τις στην αίθουσα της ε, τα κείμενα κτλ. Και αυτό το έκανα εξ ονόματος της ε, ομάδας που προεδρεύω. Και μετά είχα και δύο, ομάδες, δύο άτομα τα οποία προσέλαβα για να παρακολουθούν ε, τις εργασίες της ομάδας του 29. Επαναλαμβάνω επομένως ότι δεν έχουμε τα απαραίτητα μέσα ε, για να λειτουργήσουμε. Είχαμε πέντε διήμερα πέρυσι ας πούμε, ε, τρεις ε, συνεδριάσεις έπρεπε να τις κάνουμε μόνο μία μέρα γιατί δεν είχαμε τα τεχνικά μέσα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε πάρα πολλά θέματα τα οποία εκκρεμούν. Τώρα έφυγα από τη συνεδρίαση και είμαι σίγουρος ότι δεν θα ολοκληρώσουμε τις εργασίες μα. Έχουμε ακόμα πάρα πολλέ εκκρεμότητε έχουμε την αίσθηση ότι συνέχεια ε, κυνηγάμε τη δουλειά και δεν προλαβαίνουμε να τελειώσουμε. Και υπάρχουν θέματα τα οποία θα είναι ακόμα πιο δύσκολα, χάρη το SWIFT, διότι δεν είναι ότι δεν έχουμε ε, και όλα τα απαραίτητα μέσα για να δουλέψουμε, αλλά δεν μας δώσανε και τα, τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία θα μας επέτρεπαν να, να λειτουργήσουμε σωστά. Πρόεδρος, θα το θίξουμε το θέμα αυτό, προτείνω, αύριο το πρωί. και να, ρωτήσουμε αν ε, μπορούμε να προχωρήσουμε. Η κυρία Ένιστα, ευχαριστώ. Όπου δεν έχουμε επαρκή μέσα, έχουμε την, ε, τη δυνατότητα να μην ε, αφήνουμε τις εργασίες μας να γίνουν ολόκληρο βουνό. Και Είμαι σίγουρη ότι αυτό ισχύει και στην προκειμένη περίπτωση. Καλό λοιπόν θα είναι να το συζητήσουμε αύριο, να συζητήσουμε αύριο το πώς η ομάδα εργασίας αυτής, πώς ε, η Επιτροπή του άρθρου 29 θα τα βγάλει πέρα οικονομικά, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε και τα θέματα αρμοδιότητάς της. Το πώς μπορούν να ενισχυθούν οι δυνατότητες δράσης της, γιατί είναι απαραίτητο τέτοιες ομάδες όπου έχουν, που έχουν τέτοιες αρμοδιότητες να έχουν πιο την φωνή. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι γίνεται σήμερα, κάτι το πολύ αντιφατικό. Έχουμε αφενός το SWIFT, το οποίο έχει αποφασιστεί ουσιαστικά παρά από το γεγονός ότι θα το ψηφίσουμε, όπου περιλαμβάνονται τεράστιος όγκος προσωπικών δεδομένων που αφορούν το άτομο και τα οποία διαβιβάζονται χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει με αυτά. Και υπάρχουν αφετέρου πάρα πολλά παραδείγματα και πολύ μεγάλη άγνοια των πολιτών. Μία, αν θέλετε, διαρκής υποτίμηση του προβλήματος αυτού και πολύ το συνειδητοποιούν αυτό μόνο όταν συμβαίνει κάτι, μόνο όταν έρθουν αντιμέτωποι με την πραγματικότητα. Πραγματικά θεωρούνται ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση εις βάρος τους. Αλλά νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να συζητήσουμε στην Επιτροπή αυτή το επόμενο χρονικό διάστημα και την εισήγησή σας την κατανοώ, αν θέλετε, και την ερμηνεύω ως μια προειδοποίηση για τα πράγματα που θα μπορούσαν να συμβούν στον πολίτη τα οποία δεν τα επιθυμούμε. Θα πρέπει λοιπόν μέσω της συνθήκης της Λισαβόνας να θέσουμε πιο υψηλές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και αυτό αποτυπώνεται, από αυτή που αποτυπώνεται μάλλον, στα θεσμικά όργανα της Ένωσας. Γι' αυτό λοιπόν σας ρωτώ, αν η προστασία των δεδομένων τονωθεί ιδιαίτερα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε και να εργαστούμε σε μια τόσο μικρή ε, ομάδα εργασίας. Ποιες λοιπόν είναι οι δομές που θα πρέπει να δημιουργηθούν, να ενισχυθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αυτή τη νέα απέτηση που θέτει η Λισαβόνα. Okay. Do any other want... Μάλιστα, θέλει κανείς άλλος συνάδελφος να πάρει το λόγο. Αν μου επιτρέψετε λοιπόν να θέσω και εγώ τη δική μου ερώτηση. Καταρχάς μία παρατηρήση επιτρέψτε μου μιλήσαμε για την ανάγκη να υπάρχουν μεγαλύτερα κονδύλια για την προστασία των δεδομένων για την Επιτροπή Άρθρο 29. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι οι εταιρείε, οι επιχειρήσει φαίνεται να κατανοούν πολύ καλύτερα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία πέντε χρόνια. Όλες οι μεγάλες εταιρείε έχουν διορίσει, έχουν ε, δημιουργήσει τη θέση του υπεύθυνου προστασία δεδομένων. Κατανοούν λοιπόν πόσο σημαντική είναι αυτή και πολλέ εξ αυτών είναι πολύ σημαντικέ. Αλλά αυτό μα προκαλεί μεγάλη έκπληξη γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχη δραστηριοποίηση από τις ε, δημόσιες αρχές. Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά τι αρχέ προστασία των δεδομένων, πέρα από τους πόρους, το προπολογισμό, το προσωπικό, έχω την αίσθηση ότι ένα άλλο πρόβλημα αφορά τις περιορισμένες αρμοδιότητες εφαρμογής, κοιτώντα τι γίνεται στην Ολλανδική αντίστοιχη αρχή, υπάρχει δυνατότητα να επιβληθούν πρόστιμα, αλλά αυτά δεν έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα, καθότι είναι πολύ χαμηλά. Μπορούν ε, να παρέχουν συμβουλές και συστάσεις προς την κυβέρνηση, αλλά συχνά αγνοούνται οι συστάσεις αυτές. Θεωρείτε λοιπόν ότι θα χρειάζονταν νομικά μέσα να έχουν νομικά μέσα στη διάθεσή τους αυτές οι εθνικές αρχές προστασία των δεδομένων. Και τέλος μου προκάλεσε έκπληξη το σχόλιο σας για τα πρότυπα ISO. Ελπίζω να μην κατάλαβα σωστά γιατί τι είπατε ότι τα πρότυπα ISO αναπτύσσονται βάσει των ε, προτύπων APEC στον ΩΣΑ, δεν λαμβάνουν υπόψη δηλαδή επαρκώς τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα. Αν σωστά κατάλαβα, Προφανώς ε, θα πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό το συντομότερο δυνατόν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προτείνω η, Ευρωπαϊκή, η Επιτροπή μας να αποστείλει σχετική επιστολή, να υποβάλει ένα κοινοβουλευτικό ερώτημα, γιατί νομίζω ότι εδώ και καιρό στην Επιτροπή αυτή ζητούμε κοινά πρότυπα, συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά νομίζω ότι αν τελικά εφαρμόζονται σε εμά τα πρότυπα των αλλωνών. Αυτό δεν είναι καθόλου καλή είδηση, αν θα μπορούσατε να απαντήσετε. Ως προς το πρώτο ερώτημα, δεν μπορώ να κρίνω ένα κείμενο, εσωτερικό κείμενο του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα ήθελα όμως να πω ότι η παρακράτηση δεδομένων για μας αυτό είναι ένα θέμα ύψης της σημασίας γιατί σχετίζεται με το όλο ε, δίκτυο αφορά τις μηχανές αναζήτησης στα κοινωνικά δίκτυα. Το συζητήσαμε και προβήκαμε σε μία σύσταση πέρσι μετά από μία ακρόαση με τις βασικές, ε, βασικότερες μηχανές αναζήτησης. Το θέμα της παρακράτησης δεδομένων είναι υψίστης σημασίας διότι μπορεί να οδηγήσει στη λύθη στην ε, κοινωνία μας οι υπολογιστές έχουν τέτοιες δυνατότητες ε, μνήμης αποθήκευσης δεδομένων που ε, δεν γνωρίζουν βεβαίως την ε, λύθη, την, τη λύθη του ανθρώπινου μνημονικού. για τον άνθρωπο ε, είναι κάτι το λογικό, γιατί διαφορετικά θα κατακλυζόταν από τις επιμέρους μνήμες, ιστορικές μνήμες. Εν πάση περιπτώσει, τα δεδομένα δεν πρέπει να τα κρατάμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία. Εμείς αντιτιθέμεθα στις παρακρατήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποτανθήκαμε στις ε, μηχανές αναζήτησης λέγοντας ότι το εξάμεινο είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα αποθήκευσης δεδομένων. Συμφωνήσαμε δηλαδή για ένα μέγιστο χρονικό διάστημα έξι μηνών και σήμερα γίνονται συζητήσεις στα πλαίσια των υπευθύνων μηχανών αναζήτησης που λένε ότι ίσως οι έξι μήνες θα πρέπει να παραταθούν σε εννέα κλπ σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Ε, βεβαίως βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη στιγμή και θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ένας από τους ε, βασικούς μας εχθρούς ως προς την προστασία δεδομένων έγκυται στο ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ε, κινούνται με μία ψευδολογική λέγοντας ότι ε, είναι ενήλικοι, ενήλικες και δεν έχουν να αντιτάξουν τίποτα. Αλλά αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με την ε, πρακτική μας πορεία. Διότι η έννοια της ε, ελεύθερης, της συμφωνίας τι σημαίνει το ότι συμφωνώ με κάποιον χωρίς να προβάλλω αντιρρήσεις. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε, α, δεν έχω να κρύψω τίποτα. Ας μου παίρνουν δακτυλικά αποτυπώματα, ας με παρακολουθούν κάμερες και το καθεξής. Μα αυτό αποτελεί μεγάλη σύγχυση, διότι αθότητα δεν σημαίνει και εκφοπισμό. Δηλαδή, ε, δεν πιστεύω ε, ότι θα πρέπει να λέμε «Α, εφόσον έχω την νόμιμη σύζυγό μου μπορούν να με παρακολουθούν». Όμως εφόσον έχω μία ερωμένη δεν θέλω να με παρακολουθούν. Αυτό είναι εντελώς λανθασμένο. Σας παίρνω ένα ακραίο παράδειγμα, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει ε, δικαίωμα παρακολούθησης, δηλαδή δεν προβάλλουμε το τεκμήριο της αθωότητας για να πούμε αν μπορεί ή δεν μπορεί κάποιος να μας παρακολουθεί, δηλαδή το ζωτικό μας χώρο, το ζωτικό μου χώρο δεν θέλω να μου τον παραβιάσει κανείς χωρίς τη συγκατάθεσή μου, όποια και να είναι η κατάσταση. Αν και δεν έχω τίποτα, να, τίποτα το κακό στην συνείδησή μου. Εγώ είμαι καθηγητής πανεπιστημίου, έχω φοιτητές 19 ε, χρονών και ε, θεωρούν ότι αστειεύομαι όταν σου λέω κάτι τέτοιο. Μου λένε ότι ότι δεν τους ενοχλεί τη στιγμή που δεν έχουν τίποτα να προσάψουν στον εαυτό τους, αλλά νομίζω ότι ο προσωπικός χώρος είναι κάτι το ιερό, το οποίο δεν κάνει να βεβηλώνουμε. Επίσης τέθη ένα ερώτημα σε σχέση με τις επιπτώσεις της συνθήκης της Λισαβόνα. Βεβαίως αυτό είναι το θετικό μήνυμα το οποίο πρέπει να περάσουμε. Αλλά με τη συνθήκη της Λισαβόνας αυτή η συλλογιστική ίσως να επανεισαχθεί και ίσως θα πρέπει με τους πυλώνες να γνωρίζουμε ότι το z 29 και η, αστυνική, και η ομάδα των αστυνομικών αρχών θα πρέπει να, να μας ε, ξαναπασχολήσει. Βεβαίως από πάνω και όχι από κάτω, γι' αυτό θα πρέπει να επαγρυπνούμε έτσι ώστε ε, ίσως να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο πλαίσιο, πιο ενιαίο, αλλά εν πάση περιπτώσει τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχίσουν έτσι. Σήμερα είναι συμβολική ημέρα και μπορούμε να το πούμε. Για το SWIFT θα ήθελα να πω στο, στη νομική πτυχή του θέματος, αλλά νομίζω ότι σήμερα έχουμε συνειδητοποιήσει το εύρος του ζητήματος. Δηλαδή εργαστήκαμε επί του θέματος, μιλήσαμε με εμπειρογνώμονες, αλλά σήμερα είπα ότι συντάχθηκε μια έκθεση από εμπειρογνώμονες, μετέβησαν στις ΙΠΑ μας είπαν τι σκέφτονται για την κατάσταση και η έκθεση αυτή αρχιοθετήθηκε. Δεν ε, γνωστοποιήθηκε και μετά είχαμε μια συγκεφαλαίωση τριών σελίδων που ε, λάβαμε αφού παραπονεθήκαμε και το ζητήσαμε ε, επιμονα επίμονα τέσσερις-πέντε φορές. Μετά είχαμε ένα σχέδιο συμφωνίας και σήμερα το πρωί μας είπαν ότι έχει αρχαιοθετηθεί και αυτό. Όταν μου είπαν ότι αρχιοθετήθηκε, ε, μου είπε ευτυχώ κάποιο αν μπορείτε να το βρείτε σε αυτή την ιστοσελίδα, κάτι το οποίο είναι παράδοξο. Και τώρα μας λένε ότι η συμφωνία υπάρχει. αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς είναι η εξέλιξη του πλαισίου και υπάρχει και ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, διότι αυτή η συμφωνία είναι προσωρινή και νομίζω ότι στο μέλλον θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε η προστασία προσωπικών δεδομένων να τύχει ευνοϊκή μεταχείρισης στο μέλλον. Η ομάδα μας δεν αμφισβητεί την ίδια την έννοια δεν ε, τι θέμεθα κατά των καταχρήσεων και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, αλλά πρέπει να εγγυηθούμε και τις, ε, τις προσωπικές ελευθερίες. και στις τοπικές αυτοδιοίκησεις, στη δημόσια διοίκηση, όταν υπάρχουν διαφορές βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές θεωρήσεις ανάλογα με το κράτος μέλος. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει και μια εσωτερική εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης μιλήσατε για δυνατότητες θέσεις ισχύ, εφαρμογής του πλαισίου. Ορισμένες αρχές έχουν την δυνατότητα να προβούν σε πραγματικές ε, χρηματικές κυρώσεις και έχουν ειδικό βάρος. Άλλες διοικήσεις, δημόσιες διοικήσεις δεν έχουν αυτή την, αυτό το ειδικό βάρος. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Ε, ορισμένες υπηρεσίε έχουν υψηλά κλιμάκια πραγματογνωμοσύνης, άλλοι όχι. Εγώ δεν κατακρίνω τους μεν ή τους δε. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ αρχών. Και γι' αυτό είπα στην αρχή ότι έχω την εντύπωση ότι στο μέλλον, με, μέσα στα πλαίσια του άρθρου 29, ίσως θα πρέπει όλοι να χρησιμοποιήσουμε τα διάφορα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, διότι στην προστασία δεδομένων υπάρχει και εντάσσεται και ο παιδαγωγικός χαρακτήρας, ο χαρακτήρας της αποτελεσματικότητας θα πρέπει όμως να προβαίνουμε και σε κυρώσεις εκεί που ε, χρειάζεται και βεβαίως να υπάρχει και πραγματογνωμοσύνη. Πρέπει να συνδυάσουμε πολλά, πολλά στοιχεία και τομείς. Ναι, και θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο απότερος ρόλος μας μέσα στα πλαίσια της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ευχαριστώ. Το, το λόγο ναι, σας κύριε Σαβρέχτ. Ναι, καταρχά σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω το εξή. Ε, το τελευταίο αυτό σημείο είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα του ποια θα είναι, ποιος θα είναι ο εμπλαντικό ρόλο τη Επιτροπή Άρθρα 21 και ποιο θα είναι, ποιος θα είναι ο ρόλο του Ευρωπαίου ρεταλμένου για θέματα προσωπικών δεδομένων και θα πρέπει λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συντονιστούν τα μέτρα σε ό,τι αφορά την Europol, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών με τα τρίτα κράτη-μέλη. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο σίγουρα ε, έχει ασκηθεί μάλλον πολύ κριτική σε ό,τι αφορά την διαδικασία SWIFT. Θα ήθελα να τονίσω λοιπόν ένα θέμα ακόμη σε ό,τι αφορά την διαφάνεια στην νομοθετική διαδικασία. Νομίζω ότι αυτό αποτέλεσε ένα σαφές μήνυμα για το πώς υπάρχει στην Ευρώπη μια διαδικασία μυστικής, αν θέλετε, νομοθεσίας, την οποία δεν δεχόμαστε σε, σε καμία περίπτωση. Εδώ θα πρέπει λοιπόν να βγούμε και να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν να αποφασίζονται τέτοιοι νόμοι και να μην δημοσιεύονται, να μην ε, γίνονται γνωστοί στο ευρύ κοινό, όπου μιλάμε για ελευθερία πληροφόρησης, τίθεται και θέμα προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών και των προσωπικών δεδομένων. Αυτό που θα με ενδιέφερε τέλος είναι το εξής. Πώς θα πρέπει θετικά να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση πλέον προκειμένου να καταργηθούν οι δομές των πυλώνων και ποια είναι τα ελάχιστα πρότυπα σε ό,τι αφορά τον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων του πολίτη και θεωρώ ότι θα είχε νόημα, θα ήταν ωφέλιμο η προστασία των δεδομένων, η οποία υφίσταται, η οποία σαφώς και μπορεί να βελτιωθεί σε κάποιους ε, τομείς, αλλά έχει μια καλή βάση να αποτελέσει και τη βάση για τη συνεργασία στον τρίτο πυλώνα για την ανταλλαγή πληροφοριών στον τρίτο πυλώνα. Και ίσως ε, με την ε, συνθήκη 108 του Συμβουλίου να τεθούν κάποια πρότυπα τα οποία θα μπορούσαν να ορίσουν, αν θέλετε, και τις εξαιρέσεις, αντί να κάνουμε το αντίστροφο, όπως κάναμε ως τώρα, και να λέμε δηλαδή ότι αυτά δεν ισχύουν στο συγκεκριμένο τομέα και απλά ορίζουμε κάποιες διατάξεις ε, προστασίας για την προστασία των δεδομένων. Να δούμε λοιπόν μήπως η οδηγία για την προστασία των δεδομένων από τον πρώτο πυλώνα να μεταφερθεί και εκεί. Να δούμε δηλαδή τι γίνεται με τη συνεργασία αυτή. Και να πω και το εξή. Να μην μιλάμε για τις αρχές, για την προστασία των δεδομένων πάντα, αλλά να δούμε και τι γίνεται με τις διατάξεις για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, δηλαδή δικαστικές αποφάσεις. Να δούμε τι γίνεται με τις δικαστικές αποφάσεις. αντί να μιλάμε έτσι γενικά και αόριστα για τις αρχές αυτές. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Μία παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε, πριν σας ζητήσω να απαντήσετε. Είπατε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε το EDPS. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να ενισχύσουμε και την ομάδα εργασία ε, του άρθρου 29, διότι θα πρέπει να το συγκρίνουμε και με τα άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα επίβλεψης, ας πούμε. Ε, ας πούμε, αν έχουμε να το συγκρίνουμε με τα δίκτυα των επιθεωρητών των, ε, ε, των αγορών, θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και θα πρέπει να να δούμε πόσο ο Ευρωπαίος επόπτης προστασίας των δεδομένων θα χειριστεί το, το, σύστημα α, κοινοποίησης των παραβιάσεων ας πούμε της νομοθεσίας γιατί θα έχουμε εκατοντάδες ακόμα κοινοποίησεις παραβίασης της νομοθεσίας με τις οποίες θα πρέπει να ασχοληθείτε. Θα ήθελα πριν να απαντήσω στο ερώτημά σας, θα ήθελα να, αυτό εδώ, θα ήθελα να απαντήσω στο προηγούμενο ερώτημα για το ίζο το ΙΖΟ είναι μια ε, οργάνωση η οποία δεν είναι θεσμική αν θέλετε. Επομένως εμείς σαν ομάδα, μας, σαν ομάδα δεν ε, συμμετείχαμε ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά μας εξέπληξε το γεγονός ότι το σύνολο των εθνικών ε, οργανώσεων ΙΖΟ που είναι 200 περίπου περίπου ασχολήθηκαν με την βασική δουλειά που, ε, έκαναν, ε, που έκανε ο ΣΑ και, οι ομάδες, ε, και η ομάδα των χωρών της Αμερικής, Λατινικής Αμερικής, Βόρειας Αμερικής, Νότιας Αμερικής, Ασίας κτλ. Και θα πρέπει κάποιος παρατηρητής που θέλει να παρακολουθήσει τις ε, εργασίες ίζο μπορεί να το κάνει αλλά μέσω της ε, αντιπροσωπείας της Γαλλίας. Δεν ασκώ κριτική αλλά απλώς λέω ότι λόγω της οργάνωσης ε, και της λειτουργίας αυτής του οργανισμού δεν είναι, είναι δύσκολο, να, δεν, δεν μας επιτρέπει να συμμετάσχουμε κι εμεί ή να συνεργαστούμε, έτσι όπω θα θέλαμε τουλάχιστον. Τώρα, για το τελευταίο ερώτημα το οποίο ετέθη. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, ο κύριος Πιτσέτη και ο επόμενος πρόεδρος της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 ε, να συνεργαστούν και να μας πούνε πόσο βλέπουν να εξελίσσονται οι εργασίες ε, των δύο αυτών ομάδων για να ενταχθούν καλύτερα στην συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει το θεσμικό σταυροδρόμιο, αν θέλετε, που είναι η συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά υπάρχει ένα άλλο σταυροδρόμιο που είναι η τεχνολογία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η τεχνολογία ε, εντάσσεται και αναμειγνύεται στη δουλειά, στην καθημερινότητά μας όλο ένα ε, και ε, περισσότερο. Και θα πρέπει να ληφθεί μια σωστή απόφαση για να είμαστε αποτελεσματικοί. Και για να απαντήσω τώρα στον τελευταίο συνάδελφό σας, η προστασία προσωπικών δεδομένων είναι κάτι πολύ πιο βαρύ από αυτό το οποίο φανταζόμαστε. Γιατί θα μας επιτρέψει να διατηρούμε τις βασικές μας και τις θεμελιώδεις μας ελευθερίες σε μια κοινωνία έτσι όπως είναι αυτή σήμερα. Μπαίνουμε σε μια ψηφιακή κοινωνία. Το σύνολο της καθημερινής μας ζωής, είτε το θέλουμε είτε όχι, θα είναι σε συνεχή επαφή με αυτή την τεχνολογία. Η προστασία των δεδομένων θα μας επιτρέψει να ασκούμε την ελευθερία έκφρασης και τις άλλες θεμελιώδεις ελευθερίες σε μια κοινωνία η οποία θα έχει αλλάξει ριζικά. Εάν αυτός ο μηχανισμός δεν εξεταστεί σε υψηλό επίπεδο και λυπάμαι ας πούμε, γιατί και, στην, και, στη Γαλλία ισχύει αυτό, λυπάμαι ιδιαίτερα γιατί από τις 7 χώρες της κοινότητας μόνο οι 13 έχουν αποφασίσει να εντάξουν στο Σύνταγμα την ελευθερία ε, κάποιες ελευθερίες και πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει αυτό έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων ε, εξασφαλίζει, θα εξασφαλίσει και στο μέλλον τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λέει η Πρόεδρος, σας αξίζει να σας χειροκροτήσουμε. συνάδελφοι. Νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά στην ημερήσια διάταξη. Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης προβλέπεται για τις 5 και 4 που είναι οι ψηφοφορίες. Δεν θέλω να ξεκινήσω τις ψηφοφορίες γιατί υπάρχουν άτομα τα οποία θα έρθουν στις 5 και 4 για να πάρουν μέρος στην ψηφοφορία. Γι' αυτό προτείνω να κάνουμε ένα διάλειμμα, να επιστρέψετε όλοι εδώ στις 5 και 4 με τις κάρτες ψηφοφορίας για να ψηφίσουμε.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 Ευχαριστώ.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

Colleagues, it's almost a quarter past five. Σχεδόν πέντε και τέταρτο έχει πάει, συνάδελφοι. Okay, colleagues, can we, can we start? Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Um, well, I think I don't have all the papers here, but the first, we are going to, it's voting. Καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Θα εξετάσουμε δύο προτάσεις για προφορικά ερωτήματα. Η πρώτη, για την οποία δεν έχω απάντηση, δεν έχω συγγνώμη το κείμενο, προετοιμάστηκε με τη Συμφωνία της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών σε ό,τι αφορά την εμπορία ανθρωπίνων ανθρώπων. Μετά από συζήτηση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, Αν βλέπω ότι μου γνέφει μία από τις συζήτητρες, αν θα θέλετε πολύ πολύ σύντομα να μας παρουσιάσετε το θέμα και μετά να ψηφίσουμε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με την ε, εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνα σήμερα, νομίζω ότι το, το, το Κοινοβούλιο θα έχει πλέον και στην απόφαση σε ό,τι αφορά την εμπορία ανθρώπων. Αυτό τι σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει μια νέα πρόταση, αυτή τη φορά μια πρόταση για οδηγία, όχι για απόφαση πλαίσιο. Και αυτό θα συμβεί του χρόνου. Σήμερα συναντήθηκα δύο φορές με τους εισηγητές της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και συμφωνήσαμε να υποβληθούν ερωτήσεις προς το Συμβούλιο για το περιεχόμενο των προτάσεων αυτών. Λάβατε το κείμενο για τις ερωτήσεις αυτές και ελπίζω να τις υποστηρίξετε. Ιδανικά θα οδηγούσαν σε ψήφισμα το οποίο θα εγκριθεί στην Ολομέλεια του Στρασβούργου το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο. Το βασικό θέμα είναι αρκετά απλό. Το θέμα είναι πώς θα καταπολεμήσουμε την εμπορία ανθρώπων συνολικά. Και δεν τίθεται θέμα μόνο επί του ποινικού δικαίου, αλλά και θέμα σε ό,τι αφορά θέματα μετανάστευσης. Και θα πρέπει να δούμε τις σχετικές ε, και κατάλληλες κυρώσεις. Κατά τρίτον, θέλουμε να δούμε ποιε είναι οι συγκεκριμένες δράσεις που προγραμματίζονται, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά του Φυσικά, τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις ανάγκες των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων. Ναι, λέει η Πρόεδρος, έχουν λάβει τα μέλη τα μέλη τη εταιρεοδίση σα, άρα δεν χρειάζεται να αναπτύξετε. Να περάσουμε στην ψηφοφορία, αν θα μπορούσατε να είστε σύντομοι. Ναι, αν θα μπορούσα μόνο να θέσω μία ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Δεν ξέρω αν μου το επιτρέπετε αυτό. Ναι, αλλά με την ίδια έκκληση προς την Επιτροπή να είναι σύντομη, γιατί όλα τα μέλη είναι έτοιμα για ψηφοφορία. Είναι αυτό απαραίτητο για την ψηφοφορία. Όχι, όχι, όχι. Μπορώ να το επανέλθω σε αργότερα, σε άλλη χρονική στιγμή. Αν θα θέλατε να ψηφίσουμε την ε, ερώτηση και να θέσετε το ερώτημα αυτό στην Επιτροπή στην Ολομέλεια, εντάξει, μάλιστα. Ωραία, πολύ καλά. Οι φιλελεύθεροι ζητούν το λόγο, Ισονίν. We have a... Ναι, έχουμε ζητήσει ξεχωριστή ψηφοφορία στο 1 γάμα εάν θα μπορούσατε να λάβετε υπόψη σας το αίτημά μας. Ναι, όντως μπορούμε. Ψηφίζουμε ε, την παράγραφο 1 1Γ και ψηφίζουμε την προφορική ερώτηση στο σύνολό τη. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται μια ηλεκτρονική επιβεβαίωση, αλλά ποιοι είναι υπέρ της παραγράφου 1 1Γ. Κατά. δεν υπάρχουν, ή μία αποχή, μία αποχή πάρα πολύ καλά. Εγκρίνεται επομένως. Μπορούμε να ψηφίσουμε υπέρ της προφορικής ερώτησης στο σύνολό τη. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται, υιοθετείται και προχωρούμε και θα προχωρήσουμε προς την Ολομέλεια. Τώρα το επόμενο θέμα αφορά τα δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Η συγγήτρια είναι η Σάρα Λάτφορντ ή κάνω λάθος. Α, δεν κάνω λάθος. Καλό πράγμα είναι αυτό. Μήπως θα μπορούσατε να παρουσιάσετε εν συντομία το θέμα και μετά να ψηφίσουμε. Ναι, αλλά πριν ψηφίσουμε θα ήθελα να ακούσω από την Προεδρία και από την ε, Κομισιό την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί όπως θα θυμόσαστε αυτό είναι, μια ε, είναι ένα σχέδιο ε, και δεν, είχε, μπορούσε να υιοθετηθεί πριν από την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Ρισαβόνας. Η ερώτηση είναι πού πάμε από εδώ και πέρα. Οι υπουργοί συνεδρίασαν σήμερα στο Συμβούλιο και θα ήθελα να ξέρω τι συνέβη, διότι οποιαδήποτε όλα τα μέτρα πρέπει να επαναυποβληθούν. Έχουμε τον, τον οδικό χάρτη και θα πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει, διότι το Κοινοβούλιο θέλει να διατηρήσει τον ρυθμό μας. Θα υπάρχει πρόταση από πλευρά της Κομισιόν, θα καθυστερήσει η υποβολή της πρότασης αυτής, μία ομάδα κρατών μελών θα είναι υπεύθυνη, τι θα γίνει. Θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις από πλευρά του Συμβουλίου. Και μια και είμαστε εδώ θα ήθελα οι σκιώδεις ε, εισηγητές να μου πούνε εάν θα μπορούσαν να προσυπογράψουν την ερώτηση. Πολύ, ε, πολύ καλά, ευχαριστώ. Η Σουδική Προεδρία θα μπορούσε να απαντήσει στην ερώτηση αυτή. Ευχαριστώ. Όντως ε, συνεδρίασε το Συμβούλιο χτες και σήμερα αλλά δεν ελήφθη οποιαδήποτε απόφαση για το κατά πόσον αυτό πρόκειται να υποβληθεί σαν πρόταση πρωτοβουλίας της Κομισιόν ή θα είναι πρωτοβουλία των κρατών μελών. Πάντως και η Κομισιόν και το Συμβούλιο είναι διατεθειμένα να συνεργαστούν στενά με το Κοινοβούλιο, όμως η επίσημη απόφαση δεν ελήφθη. Μόλις ξέρουμε κάτι θα σας ενημερώσουμε. Η Σάρα. Χωρίς μικρόφωνο, η Σάρα. Αυτές οι ερωτήσεις ε, θα πρέπει να υποβληθούν κάποια στιγμή. Ζητώ επομένως ε, να υιοθετήσουμε το κείμενο αυτό εδώ, ε, λαμβάνοντας υπόψη είναι τις αγγίλες που υπάρχουν. Ε, ρωτώ επίσης πάλι τους σκιώδεις συζητητές αν θέλουν να προσυμποράψουν ε, και μια και δεν υπάρχει η δέσμευση επίσημη από πλευρά των άλλων θεσμικών οργάνων θα ήθελα τα, ερωτήματα αυτά να τεθούν και στην Ολομέλεια. Μου, είπαν, μου λένε μάλλον ότι η Κομισιόν θέλει να παρέμβει σύντομα. Ευχαριστώ. Απλώς θα ήθελα να προσθέσω κάποιες προτάσεις σε αυτά που είπε η εκπρόσωπος της Προεδρίας ο πρόεδρος της Κομισιόν θα ήθελε να υποβάλει μία πρόταση με βάση το κείμενο της 8ης Ιουλίου και όχι με βάση το συμφωνημένο κείμενο του 23 Οκτωβρίου. Δεν μπορεί να το κάνει όμως αυτό επί του παρόντος μέχρι ότου αρχίσει δηλαδή να λειτουργεί η νέα επιτροπή. Από τη στιγμή που θα αρχίσουν να ε, εργάζονται οι νέοι επιτροποί, η Κομισιόν θα υποβάλει μία πρόταση με βάση το αρχικό της κείμενο. Αυτό θα γίνει όμως το νωρίτερο αρχές Φεβρουαρίου λόγω ακριβώς των δυσκολιών που, της δύσκολης συγκυρίας, χρονικής συγκυρίας. Τώρα δεν, δεν ξέρω ε, εάν τα κράτη-μέλη θέλουν να υποβάλουν κάτι νωρίτερα. Πάντως η Κομισιόν αρχές Φεβρουαρίου έχει την θέληση αυτή να υποβάλει την πρόταση. Παρα, ε, και τις δύο ερωτήσεις προς ψηφοφορία κυρία Λάτφορντ. Ναι, γιατί όχι. Από ό,τι κατάλαβα έχουμε πρόβλημα με την Ολομέλεια του Δεκεμβρίου, άρα θα πάμε στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου και αυτό είναι λίγο λυπηρόν, αλλά... Εάν έχουμε αρκετά στοιχεία μέχρι τότε, καλό είναι. Αλλά καλό θα είναι να διατηρήσουμε την πίεση. Χάρηκα που άκουσα ότι δεν θα γίνει μια νέα μελέτη ε, αντικτύπου. Δεν χρειάζεται να γίνει καινούργια μελέτη, φαντάζομαι. Ε, τώρα βλέπω, τώρα γίνονται ξεκάθαρα τα πράγματα. Ε, αν η να υποβάλει το αρχικό κείμενο, δεν χρειάζεται να κάνει την μελέτη, γιατί μας είπαν ότι αν περάσει ένα εξάμεινο θα πρέπει να γίνει μια νέα μελέτη κτλ. Κατάλαβα όλη αυτή την ε, την συνωμοσία. Διαρωτώ με, λέει, ο πρόεδρος, ή λέει η πρόεδρος, οι διερμηνείς τι καταλαβαίνουν από όλα αυτά. Ναι, ζητώ συγγνώμη, λέει η προεδρος οι διερμηνει τι καταλαβαινουν απο ολα αυτα Λάτφορντ, δεν θα το ξανακάνω. Αλλά Τέλος πάντων, εγώ προτιμώ η Κομισιόν να κάνει την πρότασή της κανονικά, αλλά για να προχωρήσει το θέμα, σε αυτήν εδώ την, με αυτήν εδώ την ευκαιρία, θα μπορούσε μια ομάδα κρατών μελών να κάνει κάτι, να αναλάβει μια κάποια πρωτοβουλία. Καλώς λέει η Πρόεδρος. Για τις ερωτήσεις. Να ψηφίσουμε τις ερωτήσεις και μετά απο, μπορούμε να αποφασίσουμε να, αποσυ... να τις αποσύρουμε εκ των υστέρων. Θα πάρετε το λόγο πριν την ψηφοφορία. Ναι, υποστηρίζω, υποστηρίζω ερώτημα. Το ερώτημα. Νομίζω ότι όπως είπατε είναι πολύ καλό να διατηρούμε την ε, φλόγα, να διατηρήσουμε ζωντανή τη φλόγα. Και μακάρι τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν την πρόταση και να αποφασίσουν ότι πρόκειται για ένα θέμα προτεραιότητας ε, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να γνωμοδοτήσει τον πιο γρήγορα. Καλώ λέει η πρόεδρο. Ας προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, ας ψηφίσουμε τώρα και αφήνουμε την κυρία Λάντφορντ, στην κυρία Λάντφορντ και στους ε, εισηγητέ ένα κάποιο περιθώριο, αν θέλετε, λιγμόν όσον αφορά την διατύπωση. Λοιπόν, ποιοι συμφωνούν να υποβάλουμε την ερώτηση. Ποιοι είναι κατά, αποχές, πολύ ωραία. Εδώ ολοκληρώνεται η δουλειά μας για σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 9. Καλό σας βράδυ. Oh, very important. Α, όχι, όχι, όχι. Μια πάρα πολύ σοβαρή ανακοίνωση στις 6.30, στις 6.30